2006 και για το Συμβούλιο Ολοκληρωμένης Αλλιευτικής Πολιτικής. Τον προηγούμενο μήνα ο εισηγητής μας παρουσίασε τον ε, ε, Μάιο το έγγραφο εργασίας, μιλήσαμε, συζητήσαμε γι' αυτό. Αυτό που θα γίνει σήμερα είναι θα μας επεξηγήσει το σχέδιο έκθεσης ο κύριος Καντέκ λοιπόν. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ο κύριος Καντέκ θα παρέμβει και μετά θα δράσει ως πρόεδρος για 15-20 λεπτά που πρέπει να απουσιάσω για να πάω σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Ο κύριος Καντέκ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, να αφήσουμε πρώτα να μπουν οι συνεργάτες και συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν πειράζει θα αλλάξω θέση, λέει ο μελητή. Όλα είναι εντάξει. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, πρώτα απ' όλα Ήθελα να επισημάνω ότι το σχέδιο εκθεσή μου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο είναι διαθέσιμο εδώ και αρκετέ ημέρε σε όλε τι γλώσσε. Σα προτείνω λοιπόν ω ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών την 28η Σεπτεμβρίου. Το παράδειγμα κατά μία εβδομάδα. 12 ώρα το μεσημέρι. Έτσι θα έχετε περισσότερο χρόνο να υποβάλλετε τροπολογίες για αυτή την έκθεση. 28 επαναλαμβάνει. Μία εβδομάδα παραπάνω. Η πρόταση της Κομισιόν και ζητώ συγγνώμη από τους εκπροσώπους της Κομισιόν είναι απολύτως μη αποδεκτή όσο έχει. Στην εκθέση μου λοιπόν προτείνω ουσιώδεις αλλαγές που σχετίζονται και με τις τροπολογίες στον βασικό κανονισμό διάβασα καθαρά στην πρόταση της Κομισιόν τη βούληση διαφοροποίησης της αλληλευτικής ε, δραστηριότητας που ουσιαστικά ανακοινώνει έναν ε, αργό θάνατο του μοντέλου αλίας στο άρθρο 32 ουσιαστικά μας μιλάει για αλλαγή επαγγέλματος ουσιαστικά των αλλήλων με τη δημιουργία ε, επιχειρήσεων εκτός της αλληλευτικής δραστηριότητας. Προτείνω κατ' ουσίαν αλλαγή αυτού του άρθρου ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις στον τομέα της αλληλείας και να δοθούν δυνατότητες δημιουργίας προς των δραστηριοτήτων σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα. Ε, μιλάμε για την τροπολογία 88. Η παραδοσιακή και παράκτη αλλήλεια παίζει θεμελιώδο ρόλο για τους τοπικούς πληθυσμούς. Ε, η Κομισιόν θέλει να προσθέσει, να δώσει επιπλέον βοήθεια, αλλά κατά την άποψή μου αυτό είναι καλό, αλλά όχι επαρκές. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα αυτής της αλληλείας. στην 93 τροπολογία προτείνουμε κάθε κράτος μέλος να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα. Εξάλλου η παραδοσιακή και η παρακτή αλληλεία έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις θάλασσες. Γνωρίζετε τη δική μου θεωρία. Αυτό που κάνει η Κομισιόν, το να δίνει έναν νέο ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι σωστό. Γνωρίζετε την απόψή μου για το θέμα. Η παραδοσιακή και παράκτη αλία δεν είναι ίδια στη Βαλτική ή στη Βόρεια Θάλασσα ή στη Μεσόγειο. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μόνο μία νέα πρόταση προτείνω λοιπόν αυτός ο ορισμός να ε, ε, αποτελέσει κομμάτι της αρμοδιότητας των κρατών μελών και έχω σχετική τροπολογία. Επίση, η πρόταση τη Κομισιόν δεν αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα τη ευρωπαϊκή Αλία. ειδικά τη γύρανση του στόλου. Τα μισά πλοία έχουν πάνω από 30 χρόνια ηλικία Υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας επί του σκάφους και ε, σεβασμού του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προτείνω λοιπόν να επενδύσουμε στην αναδιοργάνωση και ανακαίνιση του στόλου. Το έχω καταλάβει μέσω διαφόρων εκθέσεων που έχουμε ψηφίσει και μέσω διαφόρων τροπολογιών ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία από εσά, ε, η μεγάλη πλειοψηφία από εσά δεν ήσασταν υπέρ τη ε, ανανέωση του στόλου. Το ακούω και το λαμβάνω υπόψη. Θα το συζητήσουμε φυσικά σε διάφορε ευκαιρίε μέσα των τροπολογιών που θα μου υποβάλλετε. Ωστόσο η δική μου πρόταση είναι αυτή και η δική μου άποψη. Επιπλέον, αληθεύει ότι σε ορισμένε άλλε εκθέσει, για παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, το Κοινοβούλιο έλαβε θέση υπέρ τη ανανέωση. Για παράδειγμα, μέσω μια έκθεση πρωτοβουλία για την Ατλαντική Στρατηγική, ένα άρθρο που ξέφυγε, αλλά που αναφέρεται στην ανανέωση του στόλου. Δεδομένου αυτού λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε και να δούμε μεταξύ μας πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση για αυτό το δύσκολο πρόβλημα. Ε, έχουμε παρατηρήσει στην αίθουσα σχόλια. Ίσως δεν σας είδα. Α, ίσως δεν το είδατε, αλλά εγώ το είχα γράψει και το ψηφίσατε, μάλιστα. Σε, στην Ολομέλεια. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία λοιπόν στην τροπολογία 98 έχουμε ένα νέο άρθρο που χρηματοδοτεί την καταστροφή των παλαιών πλοίων και επενδύσεις για νέα πλοίο πιο ασφαλή, πιο οικονομικά και λιγότερο ισχυρά. Φυσικά υπάρχουν φραγμοί, υπάρχουν κριτήρια. Εφόσον δεχτούμε την ανανέωση του στόλου, αυτή η ανανέωση θα γίνει με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια που δεν θα αυξήσουν τη χωρητικότητα, δεν είναι αυτός ο στόχος. Είναι, το θέμα είναι να αλλιεύουμε καλύτερα, όχι να αλλιεύουμε περισσότερο. Τώρα, μέσω των συζητήσεών μας θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη απόφαση. Αυτές οι επενδύσεις δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε αύξηση της χωρητικότητας. Το επαναλαμβάνω. Προτείνω επίσης αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο να υποστηρίξει τις επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό των πλοίων, των σκαφών, και όπως κατάλαβα συμφωνούμε σχετικά επί της αρχής ε, για να βελτιώσουμε τις ειδικές εργασίες και την ασφάλεια, την εξοικονόμηση καυσίμων και τη ρήπανση. Ειδικότερα είμαι ευνοϊκός ώστε να υποστηρίξουμε την αντικατάσταση κινητήρων χωρίς να αυξήσουμε την ισχύ των πλοίων. Ουσιαστικά θα εισάγουμε κριτήρια για μείωση της ισχύω των πλοίων. Επίση γνωρίζετε ότι αντιτίθεμε στη ριζική άμεση και αυστηρή απαγόρευση των ε, από ρηπταίων ποσοτή αλλιευμάτων. Η διακατάργησή τους είναι ενδιαφέρουσα και γενναιόδορη, αλλά σήμερα είναι δύσκολα εφικτή. Πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Προτείνω αντί για αυτήν το στόχο μιας ε, μείωσης σημαντικής και σταδιακής προ αυτών των ε, ε, απορριπτόμενων αλλιευμάτων. Επίσης, ε, λυπάμαι που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλία δεν προβλέπει καμία στήριξη για τους επαγγελματίε τη Αλία που αναγκάζονται να διακόψουν προσωρινά τις δραστηριότητε τους σε περίπτωση βιολογική ανάπαυση ε, μεγάλου οικολογικού ατυχήματος ή δυσμενών περιβαλλοντικών συνθήκων. Προτείνω λοιπόν να συμπεριλάβουμε διατάξει που θα υποστηρίζουν του επαγγελματίε κατά τη διάρκεια αυτή διακοπή τη δραστηριότητά του. Αυτό αναφέρεται στην τροπολογία 130 με ταμεία αμοιβαία βοήθεια για αντιμετώπιση τυχαίων δυσκολιών. Αυτή η διατάξη επίση μπορεί να αντισταθμίζει ε, απώλειες λόγω διαφόρων εταιρείων ή λόγω των τιμών των καυσίμων, όπω έχει συμβεί στο παρελθόν. Όπω είπα, για παράδειγμα, τυχέ. Αυξήσει ε, των καυσίμων, όχι τη λογική αύξηση των καυσίμων. Ε, μια δεύτερη διάταξη μέσω της, τροπολογία ε, της τροπολογίας 131 θα καλύπτει τις προσωρινές διακοπές όπως υπάρχει ήδη. Αυτές οι δύο προτάσεις θα επιτρέπουν στους αλληλεί να διατηρούν τις δραστηριότητές τους σε περίπτωση προσωρινής διακοπής. Η κοινωνική πτυχή της PCP είναι πολύ σημαντική προτείνουμε να ενθαρρύνουμε την επαγγελματική κατάρτιση και την είσοδο των νέων στον τομέα της ελίας. Τόσο για όσους είναι ιδιοκτήτες σκαφών, όσο, και για τους μισθωτούς. Στην τροπολογία 93 προτείνω να δίνουμε πρίμες για, ε, για την εγκατάσταση νέων αλλιέων οι οποίοι αγοράζουν ένα νέο σκάφος μόλις για πρώτη φορά. Δεν πρέπει μόνο να υποστηρίξουμε δηλαδή το στόλο αλλά και το προσωπικό πρέπει να ανανεωθεί. Πρέπει να έρθουν νέοι και να πάρουν τη σκητάλη, διότι διαφορετικά θα χαθεί η Ευρωπαϊκή Αλία. Επίση, προτείνω την εισαγωγή μια συνθήκη εξάντε για την τήρηση τη νομοθεσία όσον αφορά την εργασία των εργαζομένων στον τομέα τη Αλία, στο τροπολογία 56. Στο άρθρο 141 αναφερόμαστε στις επενδύσεις για τη διαχείριση των απορριπτόμενων ελευμάτων. Δυστυχώς ε, η πρόταση της Κομισιόν δεν ασχολείται επαρκώς με άλλους τύπους επενδύσεων απαραίτητων για την ανταγωνιστικότητα των λιμένων και των στόλων. Προτείνω λοιπόν να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή του άρθρου 41 ώστε να γίνουν επενδύσεις σε όλες τις υποδομές και σε όλους τους λιμένες που υπάρχουν. Μιλάμε για την τροπολογία 122. Το άρθρο 70 ε, για την υποστήριξη των αποθεμάτων προτείνει μειούμενη ε, διατήρηση μέχρι την κατάργησή του το 2019. Εγώ αντιτίθεμαι σε αυτή την κατάργηση και θέλω να διατηρηθεί αυτός ο σημαντικό μηχανισμός για τη ρύθμιση των αγορών και των προϊόντων αλίας. Μιλάμε για τις τροπολογίες 137 και 138. Αυτό το σύστημα, το οποίο κριτικάρουμε σήμερα, θα επιτρέψει τη διασφάλιση της πώληση των προϊόντων σε τιμή σωστή για τους παραγωγούς, για τους αλληλεί. Επίσης είμαι υπέρ της συνεργασίας μεταξύ αλλιέων και επιστημόνων. Είναι απαραίτητο να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση των ταχύτερων δυνατών το αργότερο μέχρι το 2020, εκμεταλλευόμενοι όλα τα μέσα που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Η συλλογή δεδομένων έχει σημαντικό ρόλο Και προτείνουμε λοιπόν η χρηματοδότηση ε, σε αυτό το τομέα να φτάσει στο 75%. Μιλάμε για τροπολογία 147. Όσον αφορά τι ηχθειοκαλλιέργειε, είναι σημαντικό για την βιώσιμη ανάπτυξη αυτή τη δραστηριότητα να δοθούν δυνατότητε καινοτομία, επιχειρήσεων, ε, ανθρώπινο κεφάλαιο, πρόσθεση του περιβάλλοντο και δημόσια υγεία. Επιμένω στην, εμένω στη σημασία τη ηχθειοκαλλιέργεια και πρέπει να θεωρείται ω συμπληρωματική τη αλληλεία και όχι ανταγωνιστική. Επικροτώ επίσης τις προτάσεις της Κομισιόν για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη των ε, κλασικών περιοχών αλίας. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ε, είναι θετικές για την χωροταξική ανάπτυξη των παράκτων περιοχών. Οι ενοποιημένες στρατηγικής ανάπτυξης θα βοηθηθούν από τους τοπικούς οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν τους ενδιαφερομένους. Επιθυμώ και το αναφέρω στην εκθεσή μου, ο τομέας της αλληλείας και της ηχθεοκαλλιέργειας να εκπροσωπείται με, τρο... με πλειοψηφία. Αυτή είναι η τροπολογία 134. Για να ολοκληρώσω, επανέρχομαι σε ένα σημαντικό κομμάτι, την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Προτείνει η Κομισιόν στον προϋπολογισμό 332 εκατομμύρια ευρώ από το, για το, από το 2014 έως το 2020. Αυτό είναι το τετραπλάσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού αυτής της πολιτικής. Ναι, φυσικά να είμαστε φιλοδόξοι, αλλά είναι λίγο πολύ. Ναι, η αλληλευτική πολιτική πρέπει να έχει ένα σημαντικό προπολογισμό, αλλά αυτό να μην γίνεται εις βάρος της αλληλείας και των εχθειοκαλλιεργιών. Προτείνω λοιπόν ένα πλαφόν 50% εκ μέρους της ε, στην τροπολογία E57. Ε, Πρώτον λοιπόν πλαφόν 50% της PMI. Όπως βλέπετε έχω φιλόδοξες προτάσεις για την αποτελεσματική επένδυση στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Αλίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό ως, όπως δεν πρέπει να γίνει για την αλλαγή επαγγέλματος των αλίων, αλλά να αλλάξει το μοντέλο της αλίας. Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι στην, στην ε, διάθεσή σας για να συζητήσουμε και στο μέλλον φυσικά και περιμένω τις τροπολογίες σας που δεν αμφιβάλλω θα είναι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο θέλησα να παρατείνω την προθεσμία των τροπολογιών μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφοι. Ναι. Το ξέχασα ότι ο Γκάμπριελ μου είπε να προεδρεύσω για ένα διάστημα. Η Κάρμεν, η κυρία Φράγα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ έτσι κάπως να οργανωθώ. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα και έχω ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά σε ένα ταμείο αλίας. Πρώτη αποδέκτρια θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ζητείται από τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποχρεώται να παρουσιάσει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι όπως τα κράτη-μέλη, αφού θα είναι η πρώτη η Κομισιόν, θα έπρεπε να παρουσιάσει το πρόγραμμά της, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό είναι η πρώτη δικαιούχος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βοήθεια για την ανακαίνιση του στόλου, ξέρετε ότι εγώ είμαι αντίθετη προς μια τέτοια ενίσχυση. Αν ο βασικός κανονισμός ακολουθούσε αυτά τα οποία πρότεινε η Κομισιόν που δεν πρόκειται να γίνει, θα ζητούσε κατάργηση όλων των ενισχύσεων. Δεν θα γίνει έτσι όμως και θα υπάρχει κάποια συνέχεια. Άρα πρέπει να δοθεί κάποια ενίσχυση στον στόλο. Συμφωνώ εσείς ε, λέτε ε, για την προσωρινή και για την ε, ολική πάυση. θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε επίσης να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει κάθε κράτος μέλος, σε ό,τι αφορά στρέφουμε τώρα στην ερασιτεχνική αλία ή την παραδοσιακή αλία, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλοί που αλλιεύουν στην ίδια περιοχή. Δεν θα πρέπει να αποδεκατιστεί λοιπόν. Α, τώρα συγγνώμη έπιασε και βήχας. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις Πολλές φορές στα σχέδια διαχείρισης υπάρχουν παρεκκλήσεις που επηρεάζουν την παραδοσιακή αυτή ερεστέχνικη αλία. Μπορεί να υπάρξουν διακρίσεις μεταξύ Ολλανδικών, Γαλλικών ε, σκαφών κτλ. Και στο Ταμείο υπάρχει θετική διάκριση για την ε, παραδοσιακή αλία. Πώς ορίζεται όμως κάνουμε προσπάθεια να βελτιώσουμε τον σημερινό ορισμό, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια για όλους, κατά την άποψή μου. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνενέσουμε όλοι στο να βελτιώσουμε τους κανόνες για να ισχύουν τα ίδια για όλους. Όλα τα μέσα παρέμβασης ε, θα πάψουν να ισχύουν Άρα σίγουρα αυτό πρέπει να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της περίοδου προγραμματισμού. Αυτές οι ενισχύσει όμως διατηρούνται στο 2% της μέγιστης αξίας παραγωγής. Δεν μας λέτε ποια ακριβώς θα είναι η αξία. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος και αν κάνω λάθος στο συγγνώμη, αλλά νομίζω πρέπει να το διατυπώσετε κάπως διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικο-οικονομικά μέτρα, τα συνοδευτικά μέτρα. Νομίζω ότι σε αυτό το ταμείο αλίας είναι ελάχιστα αυτά. Και μεγάλο μέρος των κοινωνικο-οικονομικών ενισχύσεων είχαν να κάνουν τον παροπλισμό. Αν θέλουμε να το διατηρήσουμε ή την ε, πάυση τέλο πάντων ε, λειτουργία, αυτέ οι βοηθείε, οι οποίε, οι ενισχύσει, οι οποίε συνδυάζονται με, την, ε, με τον παροπλισμό, τη διάλυση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύονται και με κάποιο είδου αντιστάθμιση αποζημίωση. Να έχουμε ένα ταμείο κρίσης για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, φυσικών καταστροφών κτλ. Συμφωνώ. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 72 για τη μεταποίηση των ολευτικών και γεωργικών προϊόντων, νομίζω ότι η βιομηχανία της μεταποίησης έχει μείνει εκτός, είναι η μεγάλη χαμένη και καλό θα ήταν να περιληφθεί σε κάποια νέα δεσμή στο άρθρο αυτό, στο 79. Και να πω ότι ό,τι τη διαφοροποίηση που την καταργείτε είμαι εντελώ αντίθετη. Διότι διαδραμάτισε ένα πολύ θετικό ρόλο η διαφοροποίηση και εσείς την καταργείτε εντελώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, θα καταθέσω τροπολογίες που ελπίζω να σας φανούν χρήσιμες για την έκθεση. Ευχαριστώ. Merci, euh, euh, Σας ευχαριστώ πολύ, Κάρμεν, για την παρέμβαση αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ορισμό της ε, τεχνικής αλληλεία ε, ή των ε, ενισχύσεων, ναι, πράγματι αυτό που είπατε θα μπορέσουμε να το λάβουμε υπόψη μας και να το συζητήσουμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Γιάροσλα Βαλέσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα τρία πιο σημαντικά σημεία όπως πιστεύω σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Πρώτο, σε σχέση με την τροπολογία ε, που αφορά το άρθρο 2α. Η περαιτέρω χρηματοδότηση για τον εξυγχρονισμό του στόλου χωρίς να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά τα αλλιεύματα, χωρίς αύξηση του αλλιευτικού δυναμικού των σκαφών και σε σχέση και με τους κινητήρες. Λέω εξυγχρονισμός και όχι ανανέωση. Είμαστε υπέρ του εξυγχρονισμού, αν όμω τηρηθούν οι αναγκαίοι όροι και προϋπόθεσεις και αν, οι προϋποθέσεις και αν υπάρξει και η αναγκαία ισορροπία σε σχέση με το στόλο και να μην αυξηθούν φυσικά και τα αλλιεύματα, δηλαδή η αλλιευτική προσπάθεια. Και μετά έχουμε και την ανανέωση που μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να συνεπάγεται αύξηση της αλλιευτικής προσπάθειας ενώ είμαστε εναντίον αυτής της πτυχής. Προτείνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επενδύσουμε στα σκάφη του στόλου αλλά Προτείνεται επίσης και μείωση του αριθμού σκαφών. Θα πρέπει μια άλλη κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Ένα μεγάλο μέρος του στόλου της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Στόλου, ένα μεγάλο μέρος της επιρροής που ασκείται στην Αλία, αποτελεί απειλή για τα οικοσυστήματα στη θάλασσα και όσον αφορά επίσης και την ίδια την ασφάλεια στο, ε, στις δραστηριότητες των Αλιαίων. Δεύτερον, Μία τροποποίηση του άρθρου 42 προτείνεται. Όμως θα πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, με μεγαλύτερη προσοχή, διότι δεν αντανακλώνται εδώ όλες ακριβώς οι πτυχές και οι θέσεις ε, των, του τομέα των αλλιέων στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να προβληματιστούμε για την δυνατότητα υποστήριξης ε, της εσωτερικής ε, αλληλείας, εσωτερικής πλωτής ε, ή σε λίμνε αλληλεία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς ε, αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Αφορά όμως άλλες δραστηριότητες αυτό και άλλες ανάγκες από ότι στο ανοιχτό πέλαγος ή στην θάλασσα. Πάλι πρόκειται για αλληλεία. Εδώ υπάρχουν περιορισμοί ωστόσο όσον αφορά τέτοιες δραστηριότητες μέσω του Ταμείου. Τα σκάφη αυτά δεν είναι ακριβώς, ε, ας το πω έτσι, τράτες, είναι άλλου είδους σκάφη. Και μόνο σε εσωτερικές ε, ε, πλωτές δραστηριότητες αναφέρονται και αφορά αρμοδιότητα των κρατών μελών η διαχείριση αυτού του είδους της αλίας. Αυτή η αλία έχει σαν επίπτωση τη συνέπεια ότι θα εξακολουθήσει να ελέγχεται από τα κράτη Δηλαδή τελείως διαφορετικές βάσεις για τις αποφάσεις ε, δημιουργούνται εδώ. Μετά υπάρχει και το, τη αναφορά στο άρθρο 17 και σε σχέση με τα κριτήρια για την κατανομία, των επιμερισμό αυτών των κονδυλίων, των πόρων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφείς όλες οι παράμετροι. Πρέπει να αποσαφινιστούν αυτά τα στοιχεία και κυρίως να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αφορούν το μέγεθος, τη δομή και το δυναμικό του τομέα, του αλλιευτικού τομέα στα επιμέρους κράτη-μέλη. Και πρέπει να βασιζόμαστε σε γνωστά αξιόπιστα στοιχεία γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να διεξαχθεί αντικειμενικού χαρακτήρα, αντικειμενική συζήτηση για τα, τις δραστηριότητε. δραστηριότητες. Για τι επιμέρους χώρες θα πρέπει επίσης ο, ε, ο μιλητής ε, έχει επιταχύνει υπερβολικά και του ζητείτε να επιβραδύνει λίγο το ρυθμό της παρέμβασής του. Λοιπόν, υπάρχουν δυσκολίες εδώ και όσον αφορά και τα λειτουργικά προβλήματα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Και πέρα από αυτό έχουμε και κριτήρια που για την κατανομή διαμορφώνονται ή πρέπει να διαμορφώνονται έτσι ώστε η πρόσβαση στα αυτά τα κονδύλια να μην περιορίζεται για όσους ενδιαφέρονται. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιαροσλάβ. Όπως και η συνάδελφος η Κάρμεν ε, είσαι κατά της ανανέωσης αλλά υπέρ του εξυγχρονισμού του στόλου. Και τις παρατηρήσεις αυτές μπορεί να τις συμπεριλάβεις στις τροπολογίες που θα μας στείλεις. Ε, ήθελα να απαντήσω και στην Κάρμεν μιλούσες για την κατάργηση όσον αφορά τα αποθέματα. Εντάξει, ναι, μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό. Ίσως είναι κάποιο λάθος. Έχεις δίκιο. Δίνω το λόγο τώρα στο συναδελφό μας Γκουίντο Μιλάνα. Ναι, συντομία. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και, και σε αυτή τη δουλειά έχουν επικεντρωθεί οι συζητήσει τελευταία από κάποιες απόψεις. Είναι μια προσωπική σας ερμηνεία που δεν μπορούμε να μοιραστούμε όλοι. Θεωρώ ωστόσο ότι το βασικό κομμάτι του έργου σας, βάσει του οποίου συζητάμε, είναι εξαιρετικά ωφέλιμο. Και βελτιώνει ήδη την ίδια την πρόταση της Κομισιόν, που επιτρέψτε μου να πω ήταν ανεπαρκή ε, σε σχέση με την πρόταση κανονισμού. Και το θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ε, τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τα ίδια με κοινά του βασικού κανονισμού. Ουσιαστικά η πρόταση σας αυτή θα οδηγήσει στον κανονισμό. Έτσι έχουμε απόλυτη σχέση μεταξύ τη συζήτηση για την ανακαίνιση, την ανανέωση του στόλου, τον εξυγχρονισμό του, την είσοδο των νέων, την κατάρτιση. Την ίδια λογική θα ακολουθήσουμε και στο βασικό κανονισμό. Το να ε, μελετάμε αυτά τα δύο παράλληλα είναι σημαντικό. Εγώ στον κύριο Καντέκ έδωσα τι απόψει μου για το όλο θέμα και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Δύο-τρεις ερωτήσεις ήθελα να κάνω επί τη ουσίας. Συμφωνώ με την Κάρμεν που λέει ότι πρέπει να έχουμε τον ορισμό της μικρής ε, κλίμακας και παραδοσιακής αλίας. Πρώτο επιχείρημα για αυτό πρώτος λόγος για τον οποίο δίνω αυτό το επιχείρημα. Επειδή αποδεικνύεται πολύ δύσκολο λόγω της, ε, του διαφορετικού χαρακτήρα των χωρών μας να ορίσουμε τις μικρής κλίμακας, την μικρή κλίμακα παραδοσιακή αλία, προτείνω να ορίσουμε τη βιομηχανική αλία. Ή μάλιστα να κάνουμε μια προσπάθεια να ορίσουμε τι δεν είναι παραδοσιακό. Ουσιαστικά να αντιστρέψουμε το μισογεμάτο, μισό άδειο ποτήρι. Εάν δεν καταφέρουμε να πούμε τι δεν καταφέρουμε να ορίσουμε το μισογεμάτο ποτήρι, να ορίσουμε τι δεν είναι μισογεμάτο ποτήρι. Και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό κατά τι επόμενε μέρε όταν θα δώσουμε τι ε, τροπολογίε και να σκεφτούμε και αυτό το ενδεχόμενο. Πώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να το συνδυάσουμε αυτό με την υπόθεση ισχυρή ε, περιφερειοποίηση τη όλη μεταρρύθμιση. Έχουμε αποφασίσει ότι η περιφερειοποίηση είναι ένα μοντέλο που θα ορίσει τα μελλοντικά προγράμματα μέσα στα επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε κάποιο πρότυπο όπου να προβλέπεται ένας κατάλογος χαρακτηριστικών και στο πλαίσιο αυτού του καταλόγου το περιφερειακό σύστημα η αποκεντρωμένη πτυχή της μεταρρύθμισης να μπορεί να αναφέρει και να χωρίζει σε μικρό, μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις οι τύπους αλίας, ε, παράκτια, βιομηχανική, βάσει μια σειράς ευρωπαϊκών κριτηρίων που θα εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο. Ουσιαστικά το ζήτημα της μικρής μεσαίας και μεγάλης αλίας, και μεγάλης σχετίζεται με τη δυνατότητα να σχετίζεται κάποιο ε, με τα απαραίτητα πολιτικά με τα κονδύλια για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων. Και αυτό μόνο το περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή μόνο τα κράτη-μέλη ουσιαστικά μπορούν να ασκήσουν και να εφαρμόσουν ουσιαστικά και να διαβάσουν καθαρά τον νόμο για τις δικές τους χώρες. Πιστώ ότι αυτό αυτό είναι ένα άλλο μηχανισμό επίση. Α, επίση ο μηχανισμό εξυγχρονισμού και ανανέωση. Εγώ είμαι μάλλον. Θα είμαι λίγο δραστικό για τον εξυγχρονισμό. Συμφωνούμε όλοι. Όταν αντιστοιχεί στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλεία, στη μείωση τη κατανάλωση. Ναι, για την ανανέωση είναι σαφέ κατά την απόψη μου ότι πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο ανοιχτό για την ανανέωση, για την εισαγωγή νέων στον τομέα για όσους ε, αλλάζουν τη δραστηριότητά τους σε μια πιο οικολογική δραστηριότητα. Και θα σας πω, στη χώρα μου υπάρχουν ακόμα ε, σκάφη που ονομάζουμε φερετάρε, ε, μικρά σκάφη ουσιαστικά. Και εγώ λοιπόν ε, όταν έχουμε έτσι αυτό το επιβλαβές για το περιβάλλον ε, τρόπο αλληλεία και χρησιμοποιήσουμε έναν πιο επιλεκτικό, πιο οικολογικό τρόπο, σε αυτή την περίπτωση, αν μου ζητάτε να ανανεώσω το στόλο, μπορεί να συμφωνήσω. Και εδώ δεν μπορούμε απλά να πούμε ναι ή όχι, είναι πώς υποστηρίζουμε τις διάφορες δυνατότητες που έχουμε τις διάφορες κατηγορίες, τις διαφοροποιήσεις. Δεν ξέρω χρησιμοποιούμε την ίδια διαφοροποίηση, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που ζητάμε μία επιπλέον προσπάθεια να αλλιεύουμε λιγότερο, υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί ένα σύστημα ώστε ορισμένα μεγέθη και ορισμένες δραστηριότητες θα μπορούσαν να καλύπτονται και να υποστηρίζονται επειδή συμπληρώνουν τα έσοδα των αλλιών και όχι επειδή γίνονται μια άλλη, ένα άλλο επάγγελμα. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν λίγο προσοχή στη συλλογή δεδομένων και στη χρηματοδότηση της έρευνας και γι' αυτό πιστεύω πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς. Ολοκληρώνω με μια σκέψη κατά την άποψή μου σημαντική. Όταν λέτε υπάρχει μια ερμηνεία της εξήγησης ε, του κυρίου Καντέκ δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώ, είναι προσωπική. Αλλά ο κύριο Καντέκ μα μίλησε για αλληλεί, για σκάφη, για τρόπου αλληλεία. Αναφέρθηκε στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Το μόνο που δεν μας ε, λέει ο βασικός κανονισμός είναι το ψάρι. Δεν μιλάει για το ψάρι. Δεν μιλάει για τα ψάρια. Πρέπει να ασχοληθούμε να συμπεριλάβουμε στις δράσεις, να συμπεριλάβουμε δράσεις που να επιτρέπουν στις θάλασσες να παράγουν περισσότερα ψάρια, δημιουργώντας τις συνθήκες, διότι ένα κομμάτι της ουσίας εξυπηρετεί και σε αυτό. Αυτή η πρόταση δημιουργίας ε, ε, χώρων μη αλίας, no fishing areas, δηλαδή μεγάλων ζωνών όπου θα απαγορεύεται η αλία, μετασχηματίζοντας αυτό που σήμερα προβαίνουμε σε ε, ανάπαυση, ένα χρόνο κατά τον οποίο δεν αλλιεύουμε. Να μεταφέρουμε λοιπόν αυτό το χρόνο μια αλλιεύσης σε χώρο μια αλλιεύσης. Δηλαδή να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο δίκτυο το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο μη Αυτός έτσι θα φροντίσουμε, θα ασχοληθούμε όχι μόνο με τους αλληλεί και με τα σκάφη, αλλά και με τις δυνατότητες που θα δώσουμε στη θάλασσα να αυξήσει τα ψάρια. Έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα να βγούμε από την κατάσταση όπου θεωρούμε τη θάλασσα ένα ορχείο από το οποίο εξορίσουμε ψάρια και να μπούμε σε μια νοοτροπία μέσα στην οποία θα σκεφτόμαστε, θα θεωρούμε τη θάλασσα ένα χωράφι το οποίο καλλιεργούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Έξι συναρθιμοστής του λόγου. Θα δώσω τρία λεπτά στον καθένα. Κύριε Ρόντου είστε πρώτη ομιλήτρια. Παρακαλώ να μην περνάει κανείς το τρίλεπτο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια Αλάν Καρντέκ για τη δουλειά που έκανες. Ταυτόχρονα λέω ότι πιθανότατα πολλές δυσκολίες θα έχουμε. Διαβάζοντας την έκθεσή σου, μία πρόταση με προβλημάτισε που έλεγε ότι είναι όπως και τα Χριστούγεννα δορίζει, δορίζει, αλλά από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Τώρα σοβαρά όμως και όχι ανεκδοτολογικά. Σκέφτηκες καλά αυτές τις σκέψεις πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά από αυτό το ταμείο. Φοβούμε όχι. Και τώρα για το θέμα της ανανέωσης του στόλου. Η ανανέωση του στόλου είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Εφόσον υπάρχει υπερβάλλον, υπερβολικό δυναμικό <coughs> τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί θα ήταν η προσπάθεια αυτή κατά της ανανέωσης του στόλου. Πρέπει νομίζω πλειοψηφικά να καταψηφιστεί αυτό. Το θέμα της μικρής αλίας, μικρής κλίμακας αλίας, θα έλπιζα για την έκθεση Φερέρα, θα βρίσκαμε έναν ορισμό ουσιαστικά θα τα καταφέρναμε, ίσως τα καταφέραμε. Πρέπει να βρούμε έναν ορισμό ώστε για την ιδέα αυτή του Μιλάνα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα να προχωρήσουμε. Όσο δεν έχουμε ορισμό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. <clears throat> Όσον αφορά τώρα τις ε, απόρριψη αλλιευμάτων. Όταν καταστρέφονται τέτοια παράπλευρα αλλιεύματα και ξαναρίχνουμε αυτά τα ψάρια στη θάλασσα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γίνει βιώσιμη η κατάσταση και όχι να λέμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει δυσκολία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα βρούμε λύση τόσο το καλύτερο. Εξακολουθεί το αίτημα να υπάρχει για επιδοτήσεις καυσίμων. Έχουμε τον κανόνα de minimis. Μπορεί το ε, κράτος μέλος ε, επιμέρους να εξετάζει τέτοια θέματα, αλλά όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοιες επιδοτήσεις. Δεν είναι δική μας δουλειά επιδοτήσεις καυσίμων. Τώρα, πρημοδότηση και πληρωμές ε, με πριμ για τους αλληλείς, αυτό πάλι εντάσσει στην κατηγορία από πού θα προέρθουν όλα αυτά τα πριμ. Τώρα, για το Ταμείο αλία εντάξει, αλλά για την αποθήκευση να προσέξουμε, πρέπει να καθορίσουμε ακριβώς, να ορίσουμε ακριβώς τι θα γίνεται. Είχαμε στην Γεωργία ξαφνικά την κατάσταση ότι είχαμε βουνά από βούτυρο και μ, τεράστιες λίμνες ε, γάλακτος. Πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει το ίδιο με την αλληλεία. Συνεργασία με τους αλληλευτικούς τομείς. Μόνο που είναι κρίμα ότι αμέσως την πρόταση της, ε, του Συμβουλίου την ε, έκανες δεκτή 100%. Ζητήθηκε ή δυνατόν από το 2000 μια στιγμή ή μέχρι μέχρι το 2015 ή δυνατόν, το αργότερο μέχρι το 2020 να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο αίτημα του Συμβουλίου να μην όμως τηρήσουμε όλα όσα λέει το Συμβούλιο, να αναπτύξουμε δικές μας ιδέες και όχι 100% να εφαρμόζουμε αυτά που λέει το Συμβούλιο. Θα ήθελα να έχουμε μια διαφορετική πρόταση εμείς για μας για την Ευρωβουλή. Η δατοκαλλιέργεια είναι κάτι που πρέπει να ενισχυθεί στην Ευρώπη. Να έχουμε τέτοια εξάρτηση από εισαγωγή, εισαγωγές αλλιευμάτων που δυσκολευόμαστε και πρέπει να βρούμε τα σωστά μέσα και εργαλεία να λύσουμε τα προβλήματά μας. Τώρα ένα τελευταίο σημείο. Η ολοκληρωμένη αλλιευτική θαλάσσια πολιτική αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, αυτός που δημιουργήθηκε αυτό το ταμείο και πήρε αυτή την ονομασία. Και πρέπει να διαθέτει φυσικά τέτοια κονδύλια. Και μόνο έτσι μπόρεσε να λειτουργήσει αυτό ώστε να έχουμε περισσότερα κονδύλια για την αλληλεία. Να λέμε όμως ε, ότι μπορεί να γίνει ε, ό,τι επιθυμούμε και αυτό θέτει δυ, ε, δυσκολίες. Και θα έχουμε και τροπολογίες εξάλλου που θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Λέβεν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Επισήμως δεν είμαι σκιώδης. Ο συνάδελφο Ρόλι Ρωμέβα είναι ο σκιώδη εισηγητή από την ομάδα μου. Θα ήθελα να σα δώσω όμω τι απόψει τη ομάδα των Πρασίνων. Η τροπολογία 48 του εισηγητή, η οποία λέει ότι θα πρέπει να δοθούν ε, επιδοτήσεις για ανανέωση του στόλου, είναι μια τροπολογία που θεωρούμε εντελώς απαράδεκτη. Και πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα συμφωνήσουν και αυτοί ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης δεν μπορούμε να δίνουμε τα χρήματα των φορολογουμένων για έναν στόλο που ήδη έχει ε, υπερβολική, υπερβολικά μεγάλη δυναμικότητα. Άρα θεωρούμε ότι δεν είναι απόλυτα σωστό. Και είναι και ένα διέξοδο όταν μιλάμε για την ανανέωση του στόλου υπάρχει επαρκμετάλλευση και γιατί θα πρέπει να δίνουμε επιδοτήσεις ε, μόνο στους αλλοί. Σας δώσουμε τότε και σε μικρούς ε, επαγγελματίες να αγοράσουν ένα καινούριο επαγγελματικό όχημα ή ένα μικρό μαγαζί κτλ. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε όπου διαγράφηκε στην έκθεση Αλαβράκου η έκθεση Renewal ανανέωση, και ξέρω ότι ήταν στην έκθεση από την ε, Επιτροπή Ρέτζη. Δεν υπήρξε όμως καμία χωριστή ψηφοφορία, δεν έγινε καμία ονομαστική ψηφοφορία, πέρασε και ε, συγχαρητήρια. Δεν νομίζω όμως να ξαναπεράσει ή τουλάχιστον αυτό εύχομαι. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποθηκευτική ενίσχυση, storage aid. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν θετικό. Αν υπάρχει πλεόνασμα γευμάτων που δεν μπορούν να απολυθούν στην αγορά, αυτά τα λέματα θα πρέπει να μένουν στο καλύτερο σημείο αποθήκευση. Και ποιο είναι αυτό, η θάλασσα. Είμαστε κατά λοιπόν τη αποθήκευση. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα άλλο θέμα, πιστεύω ότι τα χρήματα των φορολογημένων θα πρέπει και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των αλληλευτικών πρακτικών ώστε να είναι βιώσιμε από περιβαλλοντική πλευρά. Στηρίζουμε λοιπόν την, την ε, επιλογή πιο επιλεκτικών αληφτικών εργαλείων, ε, περιβαλλοντικά βιώσιμων ε, πρακτικών. Και οι κάμερες κλειστού κυκλώματος θα ήταν και, όλες, και όλα αυτά τα μέτρα ελέγχου πιστεύουμε ότι θα ήταν πάρα πολύ θετικά. Σε ό,τι αφορά τώρα επιδοτήσεις, μάλλον επενδύσεις όταν δεν υπάρχει αποδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ της, της δυναμικότητας και της ε, βιωσιμότητας από το κράτος μέλος δεν θα πρέπει να, δίνονται, να γίνονται επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή και όταν προσαρμόζονται στα διαθέσιμα αλλιεύματα τότε θα μπορεί να παίρνουν ενισχύσεις. Θέλουμε να αποφύγουμε να δώσουμε επενδύσεις σε ένα περιττό σκάφος που κανονικά θα έπρεπε να απομακρυνθεί, αφαιρεθεί από το στόλο, γιατί μόνο έτσι θα χρησιμοποιήσουν πέφτουν τα χρήματα των φορολογουμένων. Συμφωνούμε με αυτό που είπε η κυρία Φράγκα για τη διαφοροποίηση. Η διαγραφή αυτής της έννοια θα ήταν λάθος. Υπάρχει υπερεκμετάλλευση των αλληλευτικών δυνατοτήτων και κάποιοι προσπαθούν να βρουν άλλου είδους θέσεις εργασίας. Αν θα μπορούσε να υπάρξει διαφοροποίηση εντός του αλληλευτικού τομέα, δηλαδή να ανοίξει κάποιο ένα εστιατόριο, τον αλληλευτικό τουρισμό να ασχοληθεί, να πείσει, θα μπορούσε να είναι και κάτι εντελώς διαφορετικό και αυτό θα ήταν καλό. Το θέμα είναι η προσαρμογή της, ε, της ικανότητας στα αλληλεύματα. Και αν δεν υπάρχουν αλληλευτικές δυνατότητες, δεν θα πρέπει να, προσπαθεί, να δια, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τους άλλους σε αυτό το επάγγελμα. Ο μιλά να έφυγε, αλλά ήθελα να του πω ότι εδώ δεν μιλάμε για τα ψάρια. Όχι, δεν μιλάμε για τα ψάρια. Και αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας θα μπορούσε μεταξύ άλλων να αναλάβει το να ε, περιορίσει την αχρίαστη ταλαιπωρία και βασανισμό, αν θέλετε, και των ε, ψαριών. Δηλαδή, να βρεθούν κάποιες τεχνικές για να μην υποφέρουν πλέον τα ψάρια. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θέλω να σχολιάσω και ολοκληρώνοντα θα ήθελα να πω ότι πιστεύουμε ότι τόσο άρρηκτα είναι συνδεδεμένο όλα αυτά με την έκθεση Ρόντουστ για το βασικό κανονισμό που Θεωρούμε ότι η Επιτροπή μας θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο μήπως η προθεσμία 28, Σεπτεμβρίου είναι πάρα πολύ σύντομη. Πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει με το βασικό κανονισμό και μετά να υποβάλουμε για τη δική σας έκθεση. Αλλά, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Γιατί βάζω τώρα να τρέχει το χρονόμετρο αφού κάνετε ό,τι θέλετε και δεν τηρείτε το τρέλιο από το τέλος πάντων. Λοιπόν, σας παρακαλώ, προσπαθήστε Προσπαθήστε να τηρήσετε η κυρία Τόρβαλ. Ο κύριος Τόρβαλ, διορθώνει πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε τον Αλέν για την εκθεσή του. Συζητάμε το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό ήδη. Θα προσπαθήσω λοιπόν και εδώ και αρκετή ώρα θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Επιφανειακά φαίνεται να υπάρχει κάποια γενική συμφωνία ότι χρειαζόμαστε περισσότερα ψάρια Μόλις όμως κάψουμε λίγο κάτω από την επιφάνεια, βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Και δεν νομίζω ότι σας λέω κάτι πιο μυστικό, σας αποκαλύπτω κάποιο μυστικό. Οι διαφορές αυτές αφορούν τον εξυγχρονισμό και την αλληλευτική ικανότητα και την υπερβάλλουσα αλληλευτική ικανότητα και όταν μιλάμε για αυτή την ικανότητα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο από ό,τι συνήθως θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη διάφορες πτυχές της ικανότητας. Διότι αν δεν λάβουμε υπόψη αυτές τις διάφορες πτυχές, τότε εύκολα παίζουμε ένα παιχνίδι σημειολογίας ή καθρεφτών ή στη χειρότερη των περιπτώσεων αρχίζουμε να γινόμαστε ναι. λίγο πνευματώδεις και όχι ιδιαίτερα τίμοι για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν βελτιώσουμε τις οικολογικές επιδόσεις των κινητήρων ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερα καύσιμα, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να παραμένουν περισσότερο στη θάλασσα. Ναι, ακούγεται πολύ ωραίο, τα... οι κινητήρε των πλοίων μα να είναι πιο οικολογικοί, αλλά ουσιαστικά ω αποτέλεσμα θα είχαν περισσότερη αλήφση. Θα πρέπει να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλε τι διαφορετικέ πτυχέ του εξυγχρονισμού και τη ανανέωση και να δούμε πώ επηρεάζουν την ελληνική μα ικανότητα. Βάσει αυτού μπορώ να σας αναφέρω και ένα άλλο πρόβλημα. Εάν αφήσουμε το στόλο ως έχει στην ιδιοκτησία του οποιοδήποτε βρίσκεται εκεί στη θάλασσα, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα για τις μικρές αλληλευτικές επιχειρήσεις. Διότι δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις μεγάλες με τον ίδιο τρόπο ισότιμα στην αγορά. Θα έπρεπε λοιπόν να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το πρόβλημα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε θέματα υποδομής ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή των μικρών ελευθερικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω την ε, ηχθειοκαλλιέργειες και ούτω καθεξής αλλά προερχόμενος από μια πρωτεσταντική νοοτροπία ε, θεωρώ ότι πρέπει να τηρήσω τα χρονικά όρια. Ευχαριστώ κύριε Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαρίστω να τηρήσω το χρόνο μου, αλλά θα πρέπει αυτό να ισχύει για όλους, να μην υποφέρουν εκείνοι που θα παρεμβαίνουν ύστερα, τελευταίοι μετά τους άλλους. Δεν θα χάσω το χρόνο μου γι' αυτό. Καλωσορίζω αρκετά πράγματα από αυτά που αναφέρθηκα. Υποστηρίζω με ευχαρίστη την ιδέα για κοινού ορισμούς, κοινό ορισμό όσον αφορά τα αλλιεύματα και την αλλία, να μην χάσουμε όλο μας το χρόνο για αυτούς τους ορισμούς. Πρέπει κάτι θετικό να πετύχουμε στην έκβαση αυτής της προσπάθειας. Φαίνεται με την πρόταση του κυρίου Μιλάνα ότι έχουμε κάτι παρόμοιο σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την, τον ορισμό του δραστήριου, του ενεργού γεωργού. Ίσως με κάποια στοιχεία όσον αφορά έναν ε, ε, κλειστό αρνητικό κατάλογο. Αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα περιφερειακό πακέτο που θα εκπονήσουμε ένα αρνητικό κλειστό κατάλογο, αλλά όσον αφορά και τον τομέα της ε, αλληλείας στους ε, τομείς της. Τώρα δεν θα επισέλθω σε, θέματα του βασικού κανονισμού, κάποια θέματα έχουν ήδη καλυφθεί. Έχω όμως και εγώ κάποια μελήματα, κάποιες ανησυχίες. Το είχα αναφέρει, δεν υποστηρίζω τον ε, γενικό κανόνα για την καταστροφή απόσυρση σκαφών και την ανανέωση. Θα είναι πάρα πολύ δαπανηρό αυτό και θα απομείνουν πολύ λίγα κονδύλια με ένα τέτοιο τεράστιο το κατάλογο για την ανανέωση. Θα έκανα μία εξαίρεση εδώ όμως. Αυτό θα ήταν η προώθηση και υποστήριξη με κονδύλια επιλεγμένων εργαλείων, αλευτικών εργαλείων, δηλαδή αλευτικού εξοπλισμού. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Χαίρομαι ότι ο εισηγητής σε κάποιες τροπολογίες αναφέρεται στο θέμα του πλεονάζοντος δυναμικού, αλλά θα ήθελα να είμαστε πιο αυστηροί, να αυστηροποιήσουμε με πιο αυστηρές ε, ε, διατάξεις αυτά τώρα για την αποθήκευση ή την αντιστάθμιση ή αποζημίωση για τα καύσιμα, όλα αυτά θα πρέπει να αποφύγουμε με δημόσια κονδύλια να καλύπτονται. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου σπανίζουν αυτά τα κονδύλια και περνάμε μια οικονομική κρίση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλους ατέλειωτους καταλόγους ως ευχολόγιο. Πρέπει λοιπόν να δούμε περισσότερα, να έχουμε περισσότερα κονδύλια τα οποία θα επικεντρώνονται στη συλλογή επιστημονικών στοιχείων για την επιστημονική απόδειξη με τεκμήρια της βιωσιμότητας ε, όσον αφορά τα αλλιεύματα και την αλλιευτική προσπάθεια. Χαιρετίζω κάποιες από τις τροπολογίες για την υποστήριξη του επιχειρήν, του επιχειρηματικού πνεύμα και πάλι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί η πολυμορφοποίηση, η πολυσχηδής δραστηριότητα με πλεονάζον δυναμικό είναι κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Καλοχαιρετίζω την υποστήριξη του εισηγητή για την αηφορία και τις αηφόρες πτυχές της αλίας, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη, για παράδειγμα, και υποστήριξη της μικρής κλίμακας αλίας και βιοτεχνικής αλίας. Θα έχω κάποιες τροπολογίες που θα καταθέσω που θα συμπληρώνουν αυτές τις πτυχές. Ευχαριστούν. Τρία λεπτά και ένα δευτερόλεπτα μίλησα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούν. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, τον κύριο Καντέκ διότι πολύ συγκεκριμένα το μεσοπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο και για το κοινοτικό, κοινό ταμείο αλληλείας ε, τα συνδέει με την, τον βασικό κανονισμό και με τις προτάσεις κυρίας Ρόντος και πώς ε, με τις αρχές αυτές που θέλουμε να διαμορφώσουμε τον βασικό κανονισμό θέλουμε να πρικοδοτήσουμε τέτοιες δράσεις και πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν ωφελεί να συζητάμε για να θέλουμε ε, να τροποποιήσουμε την μέγιστη αποδοτικότητα στην στην αλία όταν δεν έχουν δυνατότητες οι αλίες μας να αγοράσουν νέο εξοπλισμό για να αλλιεύουν και υποστηρίζουμε αυτή την ενεργοποίηση για να ανανεώσουν τον αλλιευτικό τους εξοπλισμό. Και τώρα αν δεν τα προσέξουμε αυτά θα πιστοδρομήσουμε βήμα προς βήμα αλλά να δούμε τι θα γίνει με τα αλλιεύματα τα οποία θα εκφορτώνονται δεν έχουμε καν προετοιμαστεί για όλες αυτές τις πρόπτικες. Να έχουμε εγκαταστάσεις για ηχθιάλευρα, και να εμπορευόμαστε τέτοιες, ε, τέτοια προϊόντα πρέπει όλα αυτά από κοινού να μας προβληματίσουν και όταν λέμε το υπερπλεονάζον δυναμικό του αλληλευτικού στόλου ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη Κανένας δεν γνωρίζει αυτό το δυναμικό ποιο είναι. Εγώ δεν το γνωρίζω. Τουλάχιστον δεν το ξέρω για τη Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία. Ποιο είναι αυτό το πλεονάζον δυναμικό. Και όταν συζητάμε για αυτά αγαπητέ Αλάν Καντέκ, ότι θέλουμε από κοινού να εξυγχρονίσουμε το στόλο, να έχουμε νέους κινητήρες, μεγαλύτερη ασφάλεια των στόλων, ε, χρειαζόμαστε ένα νεολόγιο πρώτα, ένα μητρό. Ποια είναι αυτά τα σκάφη που έχουμε και δρούν στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα. Ποιο μήκος έχουν αυτά τα σκάφη ποιο είναι το εκτόπισμά τους η δυνατότητα να φορτώνουν σε ποιο βαθμό αλλιεύματα. Και όταν λέγεται ότι δεν χρειαζόμαστε νέο δυναμικό και όλα είναι βαίνουν κακός, ε, έχουμε παλαιότερα σκάφη τα οποία μπορούν να αποσυρθούν και νέα σκάφη που θα εισαχθούν που θα μπορούν να αλλιεύουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Ορθολογικά πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να βρούμε λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Και αν το επάγγελμα του Αλιέα θέλουμε να είναι ελκυστικό στο μέλλον για τους νέους, πρέπει αυτούς τους νέους να τους δώσουμε μια προοπτική στην Αλία Γι' αυτό χρειάζονται βέβαια ε, ψάρια. Αλλά κυρία Ρόντους, τα ψάρια δεν θα τα πετύχετε με ακόμα μεγαλύτερους περιορισμούς που θα επιβάλλονται για τα χωρικά μας ύδατα. Επιπρόσθετες λέει ζώνες προστασίας. Έχουμε την Natura 2000 Θέλουμε να έχουμε ε, τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, έχουμε στις παράκτιες περιοχές αντλίες. Έχουμε παραγωγή από την αιωλική ενέργεια, ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες ώστε η βιομάζα να διασφαλίζεται για την αηφορία της ώστε να είναι διαθέσιμη στο μέλλον. Για την υδατοκαλλιέργεια, πολύ σημαντικό σημείο αυτό ιδιωτικές επενδύσεις για τις υδατοκαλλιέργειες αλλά και για τους, ε, τα, ερευνητικά ε, όργανα ώστε να είναι βιώσιμη η υδατοκαλλιέργεια πρέπει και αυτά να υποστηριχθούν και αυτά ανήκουν στις δραστηριότητες ε, του Κοινού Ταμείου Αλίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Dziękuję Panie Przewodniczący. Streszczając Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέα για την ε, δουλειά του. Και πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη ιδίω η αρχή ότι το Ταμείο θα πρέπει να βοηθά τους αλλιές και την αλλιευτική δραστηριότητα. Αυτή είναι η βασική αρχή και συμφωνώ. Από αυτήν την αρχή πρέπει να ξεκινήσουμε. Τώρα, η μικρή κλίμακα σαλία. Η υποστήριξη της μικρής κλίμακας σαλίας είναι κάτι το απαραίτητο αν συγκρίνουμε ε, την κατάσταση με την κατάσταση της βιομηχανικής αλίας και της ε, μεγάλης κλίμακας, η μικρή κλίμακα δεν θα επιβιώσει διαφορετικά. Δεν πιστεύουμε ότι με τον εξυγχρονισμό αυξάνεται το δυναμικό η αλληλευτική ικανότητα. Αν κάποιο αγοράσει ένα άλλο αυτοκίνητο με την ε, ε, με μεγαλύτερη υποδύναμη μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα. Όχι, τόσο να αγοράσει περισσότερα καύσιμα. Αλλά ότι η υποδύναμη, η δύναμη του κινητήρα, αν παραμείνει ίδια δεν θα αυξηθεί η αλληλευτική ικανότητα. Στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για, τη... για τους κινητήρες των σκαφών. Σίγουρα αυξάνουμε την ασφάλεια όμως με τον εξυγχρονισμό. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. 45 χρονών είναι ο μέσος όρος των σκαφών στην Πολωνία. Υπάρχουν και άλλα 17 μέτρων, αλλά τέλος πάντων πρέπει να εξυγχρονίσουμε το στόλο μας, αυτό είναι σίγουρο. Ο βιομηχανικός στόλος έχει εξυγχρονιστεί. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα μικρής κλίμακας αλλιευτικά σκάφη. Δεν θα συμφωνήσω ποτέ να αναλάβουν τη δραστηριότητα της μικρής κλίμακας αλλία, αλίας σκάφη από τον βιομηχανικό στόλο. Πρέπει να προστατεύσουμε τη μικρή κλίμακα αλλία. Κάποια κράτη για να προστατεύσουν το περιβάλλον πρέπει να στηρίξουν τη μικρή κλίμακα αλίας, όχι τα μεγάλα πλοία. Σε ό,τι αφορά τι απορρίψει, η ιδέα τη αποθήκευση είναι πολύ καλή ω μέθοδος αντί των απορρίψεων, γιατί σίγουρα πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να εγκαταλείψουμε την πρακτική των απορρίψεων. Άμεσα να την εγκαταλείψουμε, χωρίς όμως να καταστρέψουμε τον αλληλευτικό τομέα. Εν γέννη λοιπόν στηρίζω την έκθεση του Άλεα. Ευχαριστώ ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρόντου, είχε ζητήσει ξανά το λόγο. 30 δευτερόλεπτα σας δίνω. να Η κυρία Ρόντου. Όχι, μόνο μια πρόταση. Θέλω να σας παρακαλέσω το EMFF σε σχέση με τον βασικό κανονισμό να το εγκρίνουμε. Γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα η δουλειά που κάνουμε εδώ αν δεν το εγκρίνουμε. ¿Cómo? ¿Es el, lo, todo lo contrario de Μπορείτε να εξηγήσετε τι είπατε. Είπατε να ψηφίσουμε αυτό. Ε, θα το δούμε στο τέλος της συζήτησης. Να ψηφίσουμε πρώτα τον βασικό κανονισμό και μετά το, ε, χρηματοοικονομικό ε, την χρηματοοικονομική πρόταση. το αντίθετο αναφέρθηκε, όχι. Εντάξει, εντάξει λοιπόν, από την Επιτροπή θα παρέμβει κάποιος. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά εξετάζει, μελετά όλε τι προτάσει του εισηγητή με μέγιστο ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή δεν θα τοποθετηθούμε ακόμα. Απλά και μόνο δύο πράγματα ήθελα να πω. Το πρώτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το φω των συζητήσεων εξακολουθεί να είναι πεισμένη ότι η πρότασή τη υπό γενικού όρου εξακολουθεί να είναι η καλή πρόταση, θετική πρόταση. Πέρα από αυτό, διατυπώθηκε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ένα συγκεκριμένο ζήτημα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα χρηματοδοτικά που θα ήθελα από πλευράς Ντομινίκ να απαντηθεί εξειδικευμένα από τον συνάδελφο. Ευχαριστώ σε τέφαρο το ρήμα της κυρίας Φράγκα για το γεγονό ότι τα ταμεία άμεση διαχείριση δεν θα αποκλειθούν σε προγραμματισμό. Πράγματι, αληθεύει αυτό. Δεν θα είναι πολυετή ο προγραμματισμό, αλλά υπόκειται στον έλεγχο τον κοινοβουλευτικό και αυτό σε αιτήσια βάση. Ενώ οι εθνικοί περιπολισμοί δεν υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο προ έγκριση, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον. Όπου να είναι θα γίνει και αυτό. Ωραία, ακούσαμε λοιπόν και την Επιτροπή. Α δώσουμε ξανά το λόγο στον κύριο Καντέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά όλους τους συναδέλφους μου για τι παρεμβάσει του, Είχα αρχίσει να απαντώ στην Κάρμεν και στον Γιάροσλαβ. Δεν έχω απαντήσει συγκεκριμένα στον ε, Γκίντο ή στην Ουλρίκε. Ίσως συναδέλφους η Ιζαμπέλα, Νίλ, νιλ και τα λοιπά. Δεν μπορώ να απαντήσω βέβαια σε όλα, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορώ αυτή τη στιγμή να σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα η ιδέα του Κίντο Μιλάνα που λέει ότι είναι δύσκολο να ορίσουμε ε, την παραδοσιακή ιερασταχνική αλία, αλλά πιο εύκολο είναι να ορίσουμε ό,τι δεν είναι παραδοσιακή αλία. Ε, ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή, σε ό,τι αφορά τώρα τη διαφοροποίηση. Δεν έχω κλείσει όλες τις πόρτες στις προτάσεις μου για την διαφοροποίηση. Δεν θα, σε δεν θα δεχτώ αυτό που λέτε, γιατί δεν αληθεύει. Ποτέ δεν έκλεισα όλες τις πόρτες. Είναι ακόμα δυνατή η διαφοροποίηση. Και Ουλρίκε, ναι, πράγματι δεν είμαι και ο Βασίλη, άσπρα γενιάδα δεν έχω, Τέλο πάντων. Εμεί συλλογικά έχουμε 6,5 δι ευρώ για αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλία. Φυσικά και έχουμε περιορισμένο προπολογισμό και οι προτάσει τι οποίε σα διατυπώνω λαμβάνουν υπόψη του περιορισμού αυτού. Θα χρειαστεί να κάνουμε επιλογέ, όπω καταλαβαίνετε και αυτό ακριβώ κάνουμε εδώ. Δεν είμαι σίγουρα και Βασίλη. το επαναλαμβάνω για την Ιζαμπέλα. Δεν μπορώ τώρα να σχολιάσω όλα τα συμμετοπέα ανέφερες. Απλά λυπούμε για το ότι ενίοτε ακολουθείται μια άκρο ιδεολογική προσέγγιση και κάποιες φορές αυτό με ενοχλεί. Βέβαια, διατυπώνεται κάποιες προτάσεις τις οποίες ε, θα χαρακτήριζαν ενδιαφέρουσες σε σχέση με αυτές που κάνω εγώ κάποιες φορές. Τον Νίλς επίσης με πολύ μεγάλη προσοχή τον άκουσα, άκουσα τις παρατηρήσεις του. Ενδιαφέρουσες ήταν, εύστοχες ήταν και τη Ζουλή ε, που και αυτή έκανε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και σε ό,τι αφορά τον Βέρνερ που μίλησε για συγκεκριμένους στόχους, πράγματι για αυτό το ταμείο προσπαθώ να δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Συγκρατώ επίσης και την παρατήρηση του Βέρνερ ότι και πολλών άλλων, ε, το λέω και το ξαναλέω, το γνωρίζετε, δεν γνωρίζουμε το δυναμικό του ευρωπαϊκού αλληλευτικού στόλου σήμερα και λυπούμε που το λέω. Αφού λοιπόν δεν γνωρίζουμε το δυναμικό, την ε, ικανότητα, την αλληλευτική, πώς θα γνωρίζουμε το πλεόνασμα αυτής. Με, λοιπόν, πολύ το λέω. Έτσι έχουν τα πράγματα, αγαπητοί συνάδελφοι. Για μια ακόμη φορά, είναι βέβαιο ότι σε ορισμένους ε, ψαρότοπου, σε κάποιες περιοχές γίνεται αλλιευτική προσπάθεια σημαντική, υπεραλίευση, αλλά δεν νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε ορίσει το δυναμικό μπορούμε να μιλήσουμε για υπερβάλλον, για πλεόνασμα δυναμικού. Τώρα, Σε ό,τι αφορά, αγαπητοί συνάδελφοι, την απόφαση θα πρέπει να λάβουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, αν θα αποφασίσουμε πριν ή μετά το βασικό κανονισμό. Τίθεται το θέμα, πράγματι. Εγώ θα σα πρότεινα να συναντηθούμε οι σκιώδει εισηγητέ και οι εισηγητέ και οι πρόεδροι και να συζητήσουμε τι ημερομηνίε για να δούμε μήπω μπορούμε να καταλήξουμε σε μία ημερομηνία για να καταλήξουμε σε μια συνεκτική πρόταση. Συμφωνείτε λοιπόν με τον Πρόεδρο να συναντήσω εγώ τους Κιώδης την επόμενη, την μεθεπόμενη εβδομάδα και να λάβουμε μια απόφαση για τις τροπολογίες, για την ημερομηνία κατάσταση των τροπολογιών. Ωραία. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόεδρο ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντέκ. Πράγματι πολύ ωραία είναι η άποψη αυτή και αυτή η πρόταση. Τρεις ομάδες διαφορετικές, ε, τρει σχολές ακούστηκαν εδώ. Τώρα για την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη συνάντηση, αλλά εκρεμεί ακόμη η προθεσμία την κατάσταση τροπολογιών. 28 Σεπτεμβρίου ήταν. Η προθεσμία δεν ισχύει αυτό πλέον και παραμένει σε κρεμότητα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Όταν το αποφασίσουμε θα σας το ανακοινώσουμε σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή όμως δεν κλείδωσε προθεσμία. Εντάξει, παραμένει ανοιχτό το θέμα. Υπάρχει ερώτηση πάνω σε αυτό? Όχι. Ευχαριστώ. Θα είναι τουλάχιστον στις 28. Το νωρίτερο 28, ίσως λίγο αργότερα. Αυτό είπα. Μπορεί να είναι στι 28, στι 38, λέει ο πρόεδρο, ή σε τρει μήνε. Δεν έχει όμως οριστικοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Είναι σε κρεμότητα. Πότε θα είναι η προθεσμία. Ναι, παρακαλώ, κύριε Πένας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με τις προθεσμίες. Την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας υπενθυμίσει κάτι που γνωρίζετε βέβαια, αλλά είναι σημαντικό. Ό,τι έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλίας δεν είναι μεμονωμένο ή απομονωμένο, αλλά εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Υπάρχουν προθεσμίες, κοινός προγραμματισμός και υπάρχει και υποχρέωση να υπάρξει συμφωνία και για τα πέντε διαρθρωτικά ταμεία σε έφθετο χρόνο, για να είναι έτοιμα για το 2014 τα ταμεία. Επομένως, απλά σας υπενθυμίζω ότι φαίνεται να έχουμε χρόνο, μεν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι από ό,τι φαίνεται ο χρόνος μας είναι πολύ λιγότερο από αυτόν που νομίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Το λαμβάνουμε υπόψη. Ξέρετε όμως ότι και εμείς ε, διαχειριζόμαστε το χρόνο μας ε, αναλόγως. Bien, pasamos al punto 12, modificación del reglamento. Περνάμε στο σημείο 12, τροποποίηση του κανονισμού 1342 για την καθιέρωση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για το βακαλάο και το... και τους στόχους ε, και τις δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται αυτά τα αποθέματα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντότς να μας εκφράσει απόψεις της και συνεχεία όποιος άλλος συνάδελφος μπορεί να λάβει το λόγο. Έχουμε και τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Παρακαλώ κυρία Ντότς, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από αρκετού μήνε, αυτή η Επιτροπή μου ανέθεσε την ευθύνη να του αναφέρω για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για τον Μπακαλιάρο. Και εγώ θέλω ιδιαίτερα να, προχωρήσουμε με αυτό. Ωστόσο, συνάντησα διάφορες αντιπροσωπείες που ενδιαφέρονται για το κείμενο και καθίσατε σαφές ευρέως ότι ενώ η προσαρμογή του σχεδίου στη, στη συνθήκη της Λισαβόνας είναι λογικός στόχος. Αυτό που χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων του μπακαλιάρου και σχέδια για πολλά είδη. Το γεγονός ότι σχεδόν τέσσερα χρόνια ε, κατά το οποία ισχύει ο κανονισμός 1342 που είχε αντικαταστήσει έναν προηγούμενο κανονισμό για την αποκατάσταση των αποθεμάτων του Μακαλιάρου και εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με την αποκατάσταση του γάδου μας αποδεικνύει ότι απέτυχαν τα σχέδια εκείνα. Στον Ιούλιο του 2012 μετά από μια συνάντηση προσωπικού της ΤΕΦΚ επισημανθήκε ότι το τρέχον σχέδιο δεν έχει την υποστήριξη των ενδιαφερομένων και θα σας αναφέρω μια πρόταση από εκείνα τα συγκεκριμένα συμπεράσματα που λέγανε ότι ένα σχέδιο που θα έχει την υποστήριξη των ενδιαφερομένων είναι πιθανότερο να επιτύχει επειδή χρειάζεται η υποστήριξή τους για την επιτυχία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα έχουμε εδώ ενδιαφερομένους που εκπροσωπούν τη Βόρειο και άλλα περιφερειακά συμβούλια, μέλη αυτής της Επιτροπής που εκπροσωπούν όχι μόνο τη βιομηχανία αλλά και τις ΜΚΟ. Και θέλουμε να ακούσουμε τα σχόλιά τους αργότερα. Αυτή ε, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια επισημαίνουν τις πρακτικές δυσκολίες του σχεδίου που συνέβαλαν σε κάποιες δυσκολίες στον τομέα της αλίας όσον αφορά την εκμετάλλευση αυτών των υδάτων συμπεριλαμβανομένων των στόλων της ε, θάλασσας Ιρλανδίας και από τη δική μου εκλογική περιφέρεια που ουσιαστικά έχουν ελάχιστο ή καθόλου ενδιαφέρον για το γαδό τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στην Κομισιόν και εργάζονται και σε περιφερειακό επίπεδο και μαζί με τι ΜΚΟ για να καταδείξουν έναν τρόπο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε την περασμένη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη υπέβαλε την τροποποιημένη τη πρόταση για το μακροπροθέσιμο σχέδιο αποκατάσταση. Και μιλώντα σε πολλού από τον τομέα αυτών, ε, ήταν ευπρόσδεκτη αυτή η πρόταση. Περιλαμβάνει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση διάφορου συστήματα πιο φιλικά προς τους γάδους. Συστήματα αλίευσης. Χθες μαζί με άλλους συναδέλφους αυτής της Επιτροπής διοργάνωσα μια συνάντηση με τη βιομηχανία για το ζήτημα των απορρίψεων με ενθάρρυνε πολύ το πλήθος των ε, μελών αυτής της Επιτροπής που παρέστησαν. Με ενθάρρυνε επίσης το γεγονός ότι η, η βιομηχανία ήταν εδώ στο Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει τις δικές της θέσεις και τις δικές της αναλύσεις απευθείας στα μέλη του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός αυτός ο τρόπος εργασίας και ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις τους και σήμερα. Έχω ήδη κάνει πολλή δουλειά όσον αφορά την προσαρμογή του προγράμματος του μακροπρόθεσμου σχεδίου για την αποκατάσταση του γάδου στη συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι θα χρειαστούμε μια γρήγορη κοινοβουλευτική διαδικασία ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε με τις ε, τροπολογίες της ε, Επιτροπής. Ε, Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ήθελα να πω ότι και καλωσορίζω τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Ζητώ συγγνώμη αν χρειάζεται να φύγω από την Επιτροπή λίγο νωρίτερα. Έχω μια ομάδα που επισκέπτεται το κοινοβούλιο σήμερα από τη δική μου εκλογική περιφέρεια στη Βορειοϊρλανδία. Και το πρόγραμμα λέει ότι πρέπει να τους μιλήσω σε περίπου 20 με 30 λεπτά. Ίσως χρειάζεται να σας εγκαταλείψω νωρίς, σας ζητώ λοιπόν συγγνώμη. Θέλω... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντό. Θα δώσω το λόγο καταρχάς ε, στο πρώτο Περιφερειακό νομοθετικό Συμβούλιο για τα Βορειοδυτικά Ήδατα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση αυτή να προσέθω και να σας προσφωνήσω παρουσιάζοντας ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή της, ε, την βορειοδυτική περιοχή των ε, ε, υδάτων στην περιφέρεια μας. Αυτό το οποίο παρουσιάζω σήμερα είναι οι ομόφωνες απόψεις ε, του Περιφερειακού Αλευτικού Συμβουλίου των βορειοδυτικών, ε, της βορειοδυτικής περιοχής όσον αφορά τον Μπακαλιάρο. Έχω ένα μικρό αριθμό διαφανειών σε σχέση με αυτό. το βορειοδυτικό ΡΑΚ έχει ε, δημιουργεί άμεσες ανησυχίες όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα και τη λειτουργικότητα του, του σχεδίου ανάκαμψης ε, του Μπακαλιάρου με την έρευνα που κάναμε καταλήξαμε σε κάποια προσωρινά μέτρα τα οποία θα πρέπει ενεργά να παρακολουθηθούν και να μπορέσουν να, να λειτουργήσουν πριν από τα τέλη αυτού του έτους. Επίσης αναπτύξαμε μια ολόκληρη μεγάλη σειρά συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών που αναπτύξαμε και έχουμε επίσης και συνέχεια που δώσαμε Μέχρι σήμερα ωστόσο θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο στοιχεία. Τα προσωρινά μέτρα τα οποία έχουν τεράστια άμεση σημασία για μας για να επιτευχθεί μια λειτουργική λύση για το σχέδιο ανάκαμψης για τα αποθέματα μπακαλιάρου. Και δεύτερον θα ήθελα πολύ σύντομα να εισαγάγω μια νέα προσέγγιση που αναπτύξαμε σε σχέση με το βορειοδυτικό ΡΑΚ για να πάψει να φθήνει ή να πάψουν να φθήνουν τα αποθέματα του βακαλιάρου. Και έχουμε την πρώτη διαφάνεια σε σχέση με αυτό. Προτού το κάνω όμως αυτό, θα ήθελα να τονίσω το ότι το βορειοδυτικό ΡΑΚ έχει <clears throat> τρία τέτοια προγράμματα ανάκαμψης. Ένα στην περιοχή 6α, δεύτερον στην Ιρλανδική θάλασσα το 7α και τρίτον το ανατολικό, τον ανατολικό διάβλο, ανατολική διόρυγα, που και αυτό πρέπει να καλυφθεί. Ο Μπάρι που θα ακολουθήσει μετά τη δική μου παρέμβαση θα τα αναφέρει αυτά επίσης εξίσου όσον αφορά τις ε, πτυχές αυτές. Μόνο κάποιες λίγες διαφάνειες έχω σε σχέση με αυτά, όμως πρέπει οπωσδήποτε να τονίσω τη σημασία αυτού του θέματος. Έχουμε μπροστά μας προσωρινά άμεσα μέσα, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λειτουργική λύση. Συνολικά πέντε άρθρα υπάρχουν στον παρόντα κανονισμό, στο σχέδιο ανάκαμψης. Το 1342 ε, του 2008 σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Το πρώτο είναι το άρθρο 9 που έχει την αυτόματη μείωση που προβλέπει 25% κατά το 1 τέταρτο δηλαδή μείωση, αυτόματη μείωση. Και σίγουρα όταν έχουμε τα αποθέματα στην περιοχή 6α θα έχουμε μηδενικό ποσοστό αλίευσης για το 2012. Αν κάποιος μπορεί να μου πει πώς μπορεί να υπάρξει μείωση κατά 25% μηδενικού ποσοστού αλίευσης δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Πραγματικά πρέπει να προσαρμοστούν, αν προσαρμοστούν αυτές οι προτάσεις δεν έχουν κανένα νόημα όπως έχουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το δεύτερο θέμα το οποίο πραγματικά έχει κρίσιμη κέρια σημασία είναι το καθεστώς αλλιευτικής προσπάθειας. Σε σχέση με αυτό το πρώτο θέλουμε να πούμε είναι ότι επειδή είχαμε αυτές τις ε, διαρκείς μειώσεις κατά 25% των αλλιευμάτων σε αυτή τη φάση πρέπει ιδιαίτερα αυτό το καθεστώς ε, για την αλλιευτική προσπάθεια στον τομέα 6α ε, στην Ιρλανδική θάλασσα δεν λειτουργεί και έχουμε εδώ πέρα μεγάλο πρόβλημα. Σε αυτή τη φάση θέλουμε να παγώσει, να υπάρξει πάγωμα της προσπάθειας και να υπάρξει ένα με υποστήριξη, με κονδύλια που θα υποστηρίζει την μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας σχέδιο. Δεύτερον, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται σε σχέση με το άρθρο 7 δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Εδώ είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Πρέπει να απλουστευτούν και πρέπει να είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένη ε, περίοδο ως διορία. Αν κάποιοι θα έχουν τέτοιες εξαιρέσεις θα πρέπει να στοχοθετήσουμε τα αποθέματα αποτελεσματικά και όταν δείτε αυτή τη διαφάνεια πρέπει να είμαστε σε θέση γοργά να έχουμε την έγκριση τέτοιων εξαιρέσεων. Ο στόχος αφορά την αλληλευτική προσπάθεια και την κατανομή των αδειών. Και εδώ πάλι η ετήσια μείωση στην αλληλευτική προσπάθεια που ήδη προανέφερα, το 25% μείωση των αλλιευμάτων πρέπει να αφαιρεθεί, να καταργηθεί, να διαγραφεί από αυτό το πλαίσιο. Και μετά το τέταρτο άρθρο αφορά τον επιμερισμό επιπρόσθετης αλλιευτικής προσπάθειας με ειδικό εξοπλισμό. Ο ίδιος ο τίτλος τα λέει όλα νομίζω και πραγματικά από πλευράς μας ε, του ΡΑΚ ε, των βορειοδυτικών ε, υδάτων της βορειοδυτικής περιοχής πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν αποτελεσματικά αυτά όσον αφορά τον στόχο που θέλαμε να πετύχουμε και πρέπει οπωσδήποτε κάποιες από τις διατάξεις, αδιατάξεις αυτές να διαγραφούν, άλλες πρέπει να πλουστευθούν και πρέπει να έχουμε συνεκτικότητα και συνάφεια με τα ε, τρέχοντα μέτρα διατήρησης, συντήρησης των αποθεμάτων. Δεν θα επισέλθω εδώ. Έχουμε πέντε προβλήματα συγκεκριμένα που πρέπει να επιληθούν άμεσα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και τέλος, όσον αφορά τις προσωρινές τροπολογίες που έχουμε, έχουμε μια ξεχωριστή έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε που είναι ε, αξιοπρόσεκτη. Υπάρχουν κυρώσεις όσον αφορά την αλλιευτική προσπάθεια σε συγκεκριμένες ημέρες ε, που δεν μπορούμε να αλλιεύουμε. Όσο λοιπόν έχουμε, ε, έχουμε και μικρότερες διαστάσεις και του εξοπλισμού και των ματιών και όταν χρησιμοποιεί α, κανείς τέτοιου είδους ε, εξοπλισμό υφίσταται κυρώσεις ε, σε σχέση με άλλους που χρησιμοποιούν ε, μεγαλύτερα μάτια ή διαφορετικό εξοπλισμό. Δεν πετυχαίνουμε λοιπόν το στόχο μας με τέτοιου είδους αρνητικές κυρώσεις. Αυτά είναι τα πέντε κυριότερα θέματα τα οποία είδαμε σε σχέση με την άμεση δραστηριοποίηση που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Έχουμε και μακροπρόθεσμα κάποιες άλλες συνιστώσεις και έχω τις τελευταίες δύο διαφάνειες για αυτά τα θέματα. Εμείς από πλευράς του Περιφερειακού ε, Συμβουλευτικού ε, Οργάνου για την βορειοδυτική αυτή περιοχή, ίσως είμαι με κάποια ιδιοτέλεια ή μεροληπτικά τοποθετούμε. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση με συγκεκριμένες συνιστώσεις, συνιστώσεις ώστε να υπάρξει ένα προσανατολισμός όσον αφορά τα αλλιεύματα, όσον αφορά την Ιρλανδική θάλασσα και την αλλιευτική προσπάθεια εκεί. Και ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το οποίο αντλήσαμε στοιχεία σε σχέση με αυτά τον Ιούνιο του 2012 Ουσιαστικά τα συμπεράσματα ποια είναι. Είναι ότι το τρέχον σύστημα όσο όπως υφίσατε με το 1342 που προανέφερα το 2008 δεν ε, εξυπηρετεί τον στόχο που έχουμε ενώπιόν μας και θέλουμε να επιτευχθεί. Αναφέρομαι μόνο για τις περιοχές ε, ε, του Μπακαλιάρου για την αλίευσή του στην περιοχή, την βορειοδυτική περιοχή. Δεν κάνω κάποια σχόλια για τη Βόρεια Θάλασσα ή για το Σκαγκεράκι ή τον την Κατεγάτη θα ήθελα να πω ότι πρέπει να υπάρξει ένας συγκεκριμένος ε, τομέας στον οποίο θα ισχύουν αυτά τα μέτρα. Αυτό πάλι είναι περιφερειοποίηση. Δεν μπορεί ένα μέτρο ισοπεδευτικά να ισχύει για διάφορες συνιστώσεις και ακόμα για τις περιοχές ε, για τον Μπακαλιάρο, για τη βορειοδυτική περιοχή ένα τέτοιο, μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί όλες τις ανάγκες των διαφορετικών περιφερειών να τις καλύψει εξίσου ικανοποιητικά. Πρέπει να διαφοροποιηθούμε, πρέπει να δούμε λοιπόν το τι θα γίνεται σε σχέση με τα αλλιεύματα στην, ε, στα βορειοδυτικά ύδατα. Είναι μεικτό πρόβλημα και μεικτών αλλιευμάτων δεν μπορούμε ισοπεδωτικά να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει σε ένα σύνθετο μεικτό ε, σχέδιο να δράσουμε. Πρέπει να δούμε τις τεχνικές πτυχές ε, και ε, του εξειδικευμένου στόλου που πρέπει να ληφθούν υπόψη, μέγεθος ψαριών κτλ. Τώρα θα θέλαμε όλα, όλες αυτές οι αρχές να εξειδικευθούν με τον καλύτερο τρόπο ταυτοποιήσαμε, εντοπίσαμε πέντε νέα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να εντάσσονται σε αυτή την προσέγγιση. Έχουμε το, τους παραπλανητικούς όρους που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Κάθε χρόνο έχουμε ε, τον καθορισμό του TAC, Total Annual Catch, δηλαδή τον Total Allowable Catch, μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα ουσιαστικά δεν είναι μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα διότι δεν ε, συνυπολογίζονται τα, οι απορρίψεις παραπλεύρων αλλιευμάτων. Εξετάζουμε, έχουμε μπροστά μας το σύνολο λοιπόν, ε, μια ε, συνολική εικόνα που θέλουμε να καθορίζει ποια θα είναι η, τα πραγματικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Και έχουμε αρκετή σημαντική επιστημονική υποστήριξη υποστήριξη σημαντική από τους επιστήμονες, από πολλούς επιστήμονες, από διάφορα κράτη-μέλη που εμπλέκονται και καταβάλουν προσπάθειες για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Είμαστε πεισμένοι ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε μια απόλυτα νέα προσέγγιση για τον τρόπο της αντιμετώπισης και διαχείρισης του μπακαλιάρου στο 6α και 7α σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε προχωρήσει σε αυτή τη φάση πιο πολύ στην ανάπτυξη ε, και εξειδίκευση του, ε, της περιοχής α σε σχέση με την 7α. Οι άλλε αρχέ και τα άλλα θέματα που εξετάζουμε ω συνιστώσει είναι ο έλεγχο τη προσπάθεια, της αλλιευτική προσπάθειας και η Επιτροπή, η Επιτροπή σας θα μπορεί να τα επαληθεύσει αυτά. Η προσπάθεια σίγουρα πιστεύουμε εμεί και μπορείτε να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, αλλά πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει. Ο έλεγχος της αλευτικής προσπάθειας με βάση τον υπολογισμό ημερών αλλιευτικής δραστηριότητας στην ανοιχτή θάλασσα δεν δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Λέμε ότι αυτό πρέπει να καταργηθεί και να υιοθετηθεί μια νέα πιο σφαιρική, πιο αποτελεσματική προσπάθεια. Εξετάζοντας τη δυνατότητα ενός συστήματος που θα βασίζεται σε συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα, πρέπει να είμαστε σε θέση να επαληθεύουμε αν και όταν αυτά που λέμε ως ε, επιχειρηματικοί κύκλοι πράγματι αλλιεύονται και ισχύουν ή όχι. Και έχουμε αναπτύξει ένα έγγραφο θέσεων, έχουμε εκπονήσει ένα έγγραφο θέσεων για το πώς μπορούν αυτές ε, οι αλληλευτικές δραστηριότητες να τεκμηριώνονται και να ελέγχονται. Και πάλι με ένα πρότυπο δεν μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες ε, με το ίδιο ικανοποιητικά. Δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί. Πρέπει να υπάρξει διεύρυνση των δραστηριοτήτων αυτών, των συνιστοσών αυτών, να έχουμε την καλύτερη συνεισφορά από τους επιστήμονες από πλευράς προτάσεων, ώστε να είμαστε το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Φυσικά έχουμε και τα θέματα των παράπλευρων αλλιευμάτων, έχουμε και τα θέματα της ε, ε, δομής της διάρθρωσης ε, του στόλου και της προσπάθειας, κάποιες ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, η κλίμακα που πρέπει να προσαρμόζεται. Έχουμε λοιπόν αυτές τις κατευθυντηρίες γραμμές. Τώρα εργαζόμαστε ώστε να εκπονηθεί μια εξειδικευμένη πρόταση που ευελπιστούμε ότι σε κάποια φάση στο μέλλον θα μπορέσουμε να προσέλθουμε στην δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να την παρουσιάσουμε, να την παρουσιάσουμε και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξίσου. Νομίζω, Πρόεδρε, με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσα αυτά που είχα να πω σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κόνη, θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ντίς από το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Βόρεια Θάλασσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τις απόψεις ε, του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βορεια Θάλασσα. Η καθημερινή μου δουλειά είναι ίδια με τους ΣΟΝ, είμαι εκπρόσωπος για την Ελία, αλλά σήμερα ομιλώ ως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τα Βυθόβια Ψάρια και είμαι ο κ. Μπαρεντέας. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Βόρειας Θαλάσσης έχει παράγει εκπονήσει πολλές συμβουλές τα τελευταία χρόνια για το σχέδιο διαχείρισης του γάδου, αναγνωρίζοντας προβλήματα και προτείνοντας βελτιώσεις. Έχει συνεργαστεί στενά με το STCF για την αξιολόγηση του σχεδίου και των επιλογών που έχουμε για αλλαγές. Η πρόταση της Κομισιόν για ενδιάμεσες διευθετήσεις όσο το εφαρμοστεί και αναπτυχθεί ένα πλήρες ε, σχέδιο για τα βυθόβια αποθέματα που ελπίζουμε το 2014 να είναι το νωρίτερο, να είναι έτοιμο, επειδή ακόμα μελετάται. Αυτή η πρόταση έχει τώρα δημοσιευτεί. Παρότι κάποιες πτυχές των ενδιάμεσων προτάσεων χρήζουν κάποιων διευκρινήσεων και παρότι ε, απομένουν τομείς στους οποίους η Κομισιόν κατά την άποψή μας θα έπρεπε να έχει βαθύνει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά η πρόταση αναγνωρίζεται ως θετική βάσει των απόψεων των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων και των STCF. Λαμβάνει υπόψη πολλές από τις λύσεις που έχουν προταθεί. Σκοπός των προτείνομενων αλλαγών είναι πρώτο να βοηθήσουν το σχέδιο να επιτύχει τους στόχους του Συμμεριζόμενος τις απόψεις του ΣΟΝ και εμείς ε, μαζί με την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλίας θεωρούμε ότι αυτό το σχέδιο δεν θα οδηγήσει στην κατάλληλο σκοπό και ο σκοπός είναι να μειώσουμε τη θνησιμότητα των αποθεμάτων γάδου. Φυσικά οι ενδιάμεσες διευθετήσεις έχουν σχεδιαστεί για να απαλύνουν τις κοινωνικο-οικονομικές πιέσεις που σχετίζονται με τις αυτόματες μειώσεις ετησίως ε, και των συνολικών επιτρεπόμενων ελευμάτων αλλά και για την αντιμετώπιση των συνεπειών στις οποίες οδηγεί το σχέδιο τεράστια αύξηση των κανονιστικών απορρίψεων. Οι ενδιάμεσες προτάσεις Επίσης ευθυγραμμίζουν τη διαδικασία για χορήγηση εξαιρέσεων για σκάφη με ελάχιστα αλλιεύματα γάδου και παρέχει ευελιξία για το Συμβούλιο και του δίνει τη δυνατότητα να παγώσει τις μειώσεις όταν είναι αντιπαραγωγικές. Βάση επιμέρους περιπτώσεων εστιάζεται λοιπόν σε μεγάλο βαθμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αλλιευτικής δραστηριότητας και κάθε αποθέματος. Παρομοίως όπου η ISIS μπορεί να παρέχει μια αναλυτική αξιολόγηση αντικαθιστά την αυτόματη 25% μείωση με μία προσέγγιση κατά περίπτωση, την οποία εμείς επικροτούμε. Επίσης, τα σκάφη που έχουν τεκμηριωθεί πλήρως για αλεία εξαιρούνται διότι καταγράφονται όλα τους τα αλλιεύματα γάδου. Αυτό τροποποιεί ένα σχέδιο διαχείρισης ε, που υπερβαίνει τους κανόνες. Θέτει TSCs και όρια προσπάθειας. Συνεπώς θα υπαχθεί σε συναπόφαση. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το τρέχον αδιέξοδο μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για θέματα αρμοδιότητας για το σχέ... μακροπρόθεσμο σχέδιο δεν βοηθά τη γρήγορη υιοθέτηση αυτών των ενδιάμεσων διευθετήσεων διότι είναι ενδιάμεσες είναι για να καλύψουν ένα κενό έως όταν αναπτύξουμε μια πλήρη συνδυασμένη προσέγγιση για την αλληλεία. Το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο λοιπόν δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην υιοθέτηση αυτών των μέτρων σε γρήγορε ταχύε διαδικασίε εφόσον είναι αυτό δυνατόν. Διαφορετικά δεν θα έχει νόημα να υλοποιήσουμε ενδιάμεσα μέτρα τα οποία δεν θα καλύψουν τα εν λόγω κενά. Τα στοιχεία του τρέχοντος σχέδιου που έχουν λειτουργήσει σε αντίθεση με τα ολικά επιτρεπόμενα λεύματα και τον έλεγχο προσπαθειών που το STCF έχει ορίσει, όλες οι διατάξεις υπό το άρθρο 13 που ενθαρρύνουν την αποφυγή των απορρίψεων και με συνεπώς λιγότερες απορρίψεις γάδου, αυτό που έχει καταστεί σαφές ε, κατά τα τελευταία χρόνια είναι ότι αυτές οι επιτυχίες του σχεδίου θα πρέπει να αναπτυχθούν η αποφυγή των γαδών και η μείωση των απορρίψεων. Για να ολοκληρώσω, το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υιοθετηθούν αυτά τα ενδιάμεσα μέτρα θεωρούμε ότι αποτελούν ένα σοβαρό μέτρο προς τα, βήμα προ τα εμπρό. λαμβάνουν υπόψη τι συμβουλέ του STSF και των ΡΑΚ και είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ε, αληθική βιομηχανία αλλά και για τα αποθέματα γάδου εφόσον υιοθετηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ποιοι θα ήθελαν το λόγο, του βουλευτέ. Κανείς μέχρι στιγμή δεν έχει το λόγο, κύριε Λόβιν. Sí, sí, perdón. Συγγνώμη, ναι. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούμε τις απόψεις των ΡΑΚ, ακούσαμε τις απόψεις τους. Μία ερώτηση έχω προς τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Ντόναχιου. Όταν αναφερόσαστε και είπατε ότι θα θέλατε να υπήρχε ένα συνολικό επιτρεπτό αλίευμα, total allowable catch, συνολικό, σφαιρικό, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιμέρους τμήματα σε αυτό το ε, μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα. Επεξηγήσε μας ε, γιατί είναι λάθος ο υπολογισμός ο σημερινός αυτός και πρέπει να ε, διορθωθεί. Για να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα, αυτό που λέτε είναι ότι πιστεύετε ότι η σημερινή πρόταση για τον ευθυγραμμισμό του κανονισμού αυτού δεν επαρκεί. Πρέπει να τροποποιηθεί λέτε και να αλλάξει αμέσως. Αυτό είναι αυτό το οποίο μας λέτε έτσι για να είναι σαφή τα πράγματα. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ κυρία Λόβεν. Ο κύριος Κούν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και τους δύο εισηγητές ε, για από τα ε, για τις ε, παρουσιάσεις των θέσεών τους. Οι αλληλείς είναι οι πρώτοι που το βλέπουν και το παρατηρούν όταν σε κάποιο αλλίευμα δεν πάνε τα πράγματα καλά. Κάνουν μεγαλύτερες δαπάνες για το αλλίευμα ενώ έχουν μικρότερο αλλίευμα τελικά παρόλες τις αυξημένες δαπάνες. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι ποιες επιστημονικές μελέτες είχατε που αντλήσατε ακριβώς για τα θέματα του μπακαλιάρου και τα αποθέματά του και όσον αφορά τα αλλιεύματα και τα οικοσυστήματα του Μπακαλιάρου στη Βόρεια Θάλασσα και στη Δυτική Σκοτία και όλα αυτά τα οποία, ε, εντάξει, της, ε, το ράκ της Βόρειας Θάλασσας για τις ε, διάφορες χρονιές μπορεί στατιστικά να υπολογίσει κανείς και να δει σε πόσα χρόνια, τόσα χρόνια θα, είναι, θα έχει ενηλικιωθεί ένα ψάρι και τότε θα έχει αποκατασταθεί η ισορροπία των αλλιευμάτων. Σε τι οφείλεται αυτή η κατάσταση. Ίσως υπάρχει πρόβλημα με τα αυγά των ψαριών που δεν μπορούν να γονιμοποιηθούν λόγω κάποιας μόλυνσης ή επιμόλυνσης ή τις πρώτες ε, εβδομάδες ε, δημιουργούνται προβλήματα για αυτό το γόνο και μετά έτσι με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται η συνολική βιομάζα και μπορούν με αυτούς τους υπολογισμούς στο τέλος τέλος να υπολογιστούν ποια είναι τα μεγέθη που μπορούν να αλλιεύονται με την αηφορία, για να υπάρχει αηφορία, αηφόρος αλία. Θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες επεξηγήσεις. Είναι πολύ ανησυχητικό αν ένα τόσο σημαντικό ψάρι για τη διατροφή μας όπως ο μπακαλιάρος να βρίσκεται σε τόσο αρνητική κατάσταση, σε τόσο κακή θέση. Πώς μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη και βελτίωση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ο κύριος Ντόναχιου πάλι παρακαλώ να απαντήσει. Thank uh, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις δύο ερωτήσεις που νομίζω, πιστεύω ότι μπορώ να απαντήσω εγώ ίδιος. Ιδιαίτερα σε αφορά για τον κανονισμό για τα τάξ ε, και το τι πρέπει να γίνει. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Αν δούμε τον Μπακαλιάρο στην βορειοδυτική και δυτική Σκοτία, περιοχή 6α, Εφέτος υπήρχε μηδενικό ποσοστό για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα. Όμως έχουμε και απορριπτόμενα αλιεύματα. Έχουμε τεράστιο αριθμό λοιπόν αλλιευμάτων που απορρίπτονται στην θάλασσα. Αυτό που λέμε με άλλα λόγια εμείς ποιο είναι. Λέμε λένε να μην, να μην ε, ε συνυπολογίζονται τα α, αλλιεύματα αυτά. Να έχουμε μια νέα προσέγγιση. Η περιοχή 6α έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις άλλες περιοχές. Έχουμε το πρόβλημα για τον μπακαλιάρο που είναι το πρόβλημα των, απορριπτε, από, των αλλιευμάτων που απορρίπτονται. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα της μείωσης, το θέμα της μείωσης της θνησιμότητας των ε, ε, ηχθείων αυτών. Πρέπει να πάρουμε μια συνολική εικόνα, να καθοριστεί η εθνισμότητα, ε, η η αυτών των ε, ε, ψαριών και να έχουμε ανάλογη προσαρμογή αντί να έχουμε ένα μηδενικό συνολικό αλίευμα και να έχουμε από την άλλη πλευρά και το πρόβλημα των απορριπτόμενων αλιευμάτων. Πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Αυτή είναι μια συνολικά νέα προσέγγιση, εκβάθρων, ριζικά νέα προσέγγιση. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει. Αν δεν το κάνουμε δεν θα μειωθεί η θνησιμότητα των ε, ηχθείων. Η ιδέα μας ήταν ότι από τη σημερινή κατάσταση, από τη σημερινή θνησιμότητα των ηχθείων που είναι πολύ υψηλή, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια θνησιμότητα που θα είναι βιώσιμη για τον μπακαλιάρο. Αυτό θα μας έδινε τι ε, επιτρεπόμενα αλλιεύματα συνολικά κάποιων χιλιάδων τόνων ετήσια και όχι μηδενικά αλλιεύματα και όχι μόνο αυτό αλλά θα εντάσαμε, θα πρέπει να εντάξουμε σε αυτή την πρόταση και άλλα στοιχεία. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία πρέπει να είμαστε σε θέση να επαληθεύουμε το τι θα γίνεται. Αν καθοριστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πολυσχηδώς. Αυτό εκπονήσαμε και αυτό αναπτύξαμε στις συνιστώσεις του για το ΡΑΚ. Έχουμε εκπονήσει ένα συγκεκριμένο περιφερειακό έγγραφο, το οποίο βασίζεται σε αυτά τα τεκμήρια, τα επιστημονικά, για την αλλιευτική προσπάθεια. Χαίρομαι που ρωτήσατε, που θέσατε αυτό το ερώτημα. Είναι μια απόλυτα νέα προσέγγιση αυτή. Εμείς είμαστε πεισμένοι ότι στη βορειοδυτική περιοχή και δεν είναι μόνο η βιομηχανική κύκλη, η επιχειρηματική κύκλη, αυτό είναι η συνολική άποψη. Αυτό είναι εκείνο που θα καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αναφέρομαι στα αλλιεύματα στις, ε, της βορειοδυτικής περιοχής του Μπακαλιάρου. Για τη δεύτερη παρατήρηση που κάνατε, που είναι εξίσου σημαντική, Απαντώ, ναι, μάλιστα, υπέβαλα δύο σενάρια εγώ εδώ. Ε, το βορειοδυτικό ρακ θέλουμε να πετύχουμε ότι τα αλλιεύματα του μπακαλιάρου θα αντιμετωπιστούν στα προβλήματά τους που είναι τεράστια και θα τα αντιμετωπίζουμε και του χρόνου να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε με ένα, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τις επόμενες, τους επόμενους τρεις ή τέσσερις μήνες ε, να προσαρμόσουμε τις προτάσεις και να κάνουμε μια νέα προσέγγιση, εκβάθρον νέα προσέγγιση για την αποκατάσταση των αλευμάτων μπακαλιάρου. Διότι αυτό που και για τη Βόρεια ε, Θάλασσα, το, παρόν σύστημα, το παρόν σχέδιο δεν είναι δόκιμο, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και δεν θα μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία θα συνεχιστούν και του χρόνου. Ελπίζω Πρόεδρε ότι μπόρεσα να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Sí, señor, señor Δεν θα πω στις λεπτομέρειες, αλλά θα αρχιστώ να πω ότι από την εμπειρία μας και στο παρελθόν και σήμερα απλά και μόνο το γεγονός ότι συναντιόμαστε με τους ενδιαφερόμενους και τους εκπροσώπους για να μας πούν τις απόψεις τους είναι σημαντικό και ίσως θα πρέπει να το κάνουμε συχνότερα για να επαναλάβω αυτό που είπα χθε τα μέλη του Κοινοβουλίου μπορούν να συζητάνε το ίδιο το Συμβούλιο και η Κομισιόν αλλά αυτοί θέλουν βιώσιμη αλληλεία πιστεύω η βιωσιμότητα χαρακτήριζε όλα τους τα σχόλια και θα πρέπει να τα αποκριθούμε θετικά στα αιτήματά τους για κάποια μέτρα ενδιάμεσα που θα πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τα πέντε άρθρα που αφορούν τον τομέα 6α, 7α και 7d. Δεν είναι μόνο ζήτημα υποστήριξής τους. Είναι κοινή λογική, πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Το πιο απλό είναι να τα αφήσουμε όλα να κυλήσουν μόνα τους. Εγώ Πιστεύω ότι ναι, η συναπόφαση θα επηρεάσει τα πράγματα, αλλά εμεί θέλουμε το οικοσύστημα και η βιωσιμότητα να αποτελέσουν τον πυρήνα όλων των συστάσεων. Και πιστεύω έτσι θα γίνει βάσει των απόψεων της, ε, του τομέα ο κ. Δίε. Ευχαριστώ. Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τι επιστημονική υποστήριξη υπάρχει για τις συμβουλές που παρέχει το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβουλίο. Η ομάδα εργασίας για, για τη βυθοβιαλία ε, έχει επιστήμονε που συμμετέχουν σε όλες τις συναντήσεις. Πολύ ωφέλιμο για να μας βοηθήσουν στον προβληματισμό μας και στο έργο μας. Επίσης έχουμε εξυπηρήσει τις νέες ευκαιρίες που έχει ανοίξει το STCF για συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους ε, συμμετέχουμε και σε ορισμένες συνεδρίες σημαντικές του ISIS ε, όπου εξετάζονται συγκεκριμένα αποθέματα, δεδομένα και αξιολογείται οι αξιολογούνται οι προσπαθίες του. Επίσης ε, κάναμε έναν εξαιρετικό διάλογο με το ISIS για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεδομένων επιστημονικών. Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι έχουμε έναν εξαιρετικό διάλογο με τους επιστήμονες αυτή τη στιγμή που τροφοδοτεί το έργο μας. Αυτό δεν αναφέρεται πάντα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, είχαμε ένα ακραίο παράδειγμα το περασμένο Σαββατοκυριακό όπου μια γνωστή εφημερίδα η Sunday Times υποστήριξε ότι μένουν μόνο 100 ενήλικες γάδι στη Βόρειο Θάλασσα. Ουσιαστικά ο πραγματικός αριθμός είναι 21 εκατομμύρια το οποίο δείχνει την παρερμηνία που μπορεί να προκύψει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε τόσο περίπλοκα ζητήματα. Σε γενικέ γραμμέ, ε, όσον αφορά την ανάπτυξη αποθεμάτων στη Βόρειο Θάλασσα, από μια χαμηλή βάση η βιομάζα αυξάνεται έξι χρόνια διαρκώ. Κινούμαστε λοιπόν προ τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη βιομάζα. Παρότι είχαμε ξεκινήσει από χαμηλή βάση και παρότι είναι υψηλή η θνησιμότητα. Η θνησιμότητα θα έχει μειωθεί ακόμη και περισσότερο εάν είχαμε βρει μια λύση για το ζήτημα των απορρίψεων. Γι' αυτό το λόγο συμφωνούμε με αυτές τις ενδιάμεσες προτάσεις, διότι ενθαρρύνουν δυνάμει του άρθρου 13 τα μέτρα αποφυγής γάδων που πιστεύουμε θα βοηθήσουν στη μείωση των απορρίψεων. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε. Αυτό περνάμε στο επόμενο σημείο αν συμφωνείτε. Συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πήρε τον λόγο. Έχει τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Thanks, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Γνωμοδιωτικών Συμβουλίων για τις παρουσιάσεις τους. Βρεθήκαμε σήμερα σε μια κατάσταση όπου οι εκπρόσωποι του τομέα έχουν ήδη προβλέψει το περιεχόμενο της πρότασης τροποποίησης του, ετής, του πολίτου σχεδίου που υιοθέτησε η Κομισιόν στις 12 του περασμένου Σεπτεμβρίου. Και εμείς λοιπόν επικυρώνουμε τη διαθεσιμότητά μας να παρουσιάσουμε το περιεχόμενο του νέου σχεδίου των νέων τροπολογιών σε σύντομο χρονικό διάστημα και υποστηρίζουμε ότι θα θέλαμε επίση να δοθούν κίνητρα για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε αυτή η τροποποίηση να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι σημείωσα τις αναφορές που έγιναν από το εκπροσώπους του τομέα πόσο σπουδαίο είναι να διασφαλίσουμε βιώσιμη αλληλεία για το γάδο. Και το γεγονός ότι έγινε αναφορά στο στόχο ε, διακοπής του κύκλου μείωσης του γάδου και αυτός είναι ένας στόχος του σχεδίου δράσεων. αληθεύει ότι η αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής κατέδειξε το γεγονός ότι προς το παρόν το σχέδιο δεν επιτυγχάνει τους στόχους του. Αληθεύει επίσης ότι αυτό γίνεται διότι δεν υλοποιούνται ακόμα όλα τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο. Δεν ήταν δυνατό. Υπογραμμίζω ότι έγινε συγκεκριμένα αναφορά από τους εκπρόσωπους του τομέα στο ότι πρέπει να συνεχιστεί να γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να αναγνωριστούν και να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα που επιτρέπουν την αποφυγή του αλίας γαδού. Δεδομένων αυτών αληθεύει επίση ότι η αξιολόγηση τη Επιστημονική Επίτροπή και το αίτημα του τομέα αλλά και των εθνικών διοικήσεων μας οδήγησαν να προσδιορίσουμε ορισμένες αδυναμίες του σχεδίου. Αυτές οι δυναμίες, οι δυσκολίες, οι υλοποιήσεις είναι εκείνες που η Κομισιόν προτείνει με την πρότασή της να επιλύσει. Όπως υπογράμισα, η νέα πρόταση θα είναι μια πρόταση αποκλειστικά με προσωρινά μέτρα. Δεν είναι ένα πραγματικό νέο σχέδιο. Για το νέο σχέδιο η γίνεται μελέτη από την Επιστημονική Επιτροπή και από του επιστημονέ μα και ελπίζουμε να έχουμε μια πρόταση στο, σύντομο, στο προσχές μέλλον. Αποσύρω λοιπόν το αίτημα για. Ήθελα συγγνώμη, να επαναλάβω το αίτημα για μια γρήγορη συζήτηση τη νέα πρόταση τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο στη σήμερα συντάξη, το 13. Τεχνικά μέτρα ελέγχου τροποποίηση του κανονισμού 850-98 και του 1342-2008. Μια πρώτη παρουσίαση αυτών των μέτρων, το σχέδιο, έκθεσης, ε, ε, το, σχέδιο πρότασης από πλευρά της Επιτροπής. Ποιος θέλει να λάβει τον λόγο, εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προτού εισαγάγω αυτή την πρόταση για τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Σκάγκερακ, θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για αυτή την πρόταση, για να κατανοηθεί σωστά. Είναι μια σχετικά μικρή περιοχή το Σκάγκερακ. Έχει τα ύδατα όμως που συμπεριλαμβάνει της Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας. Πολύ παραδοσιακοί αλήθεια στο Σκάγκερακ περνούν, ξεπερνούν αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, τα σύνορα μεταξύ χωρικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Μέχρι σήμερα διευκολυνόταν αυτό. Είχαμε τη συμφωνία, το πλαίσιο συμφωνίας Σκάγκερακ, όπου σκάφη της Σουηδίας και Δανίας επιτρεπόταν να αλλιεύουν μέχρι και τέσσερα μίλια από την νορβηγική ακτή ενώ παρέμεναν υπό τα πλαίσια της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όπως ίσως γνωρίζετε, κατάργησε αυτή τη συμφωνία, την ήρε η Νορβηγία. Έτσι από την 8η Αυγούστου 2012 πλέον, σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις για την ε, παράκτη αλία όσον αφορά την περιοχή του Σκάγκερακ. Έχουμε λοιπόν διαφορετική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Νορβηγία. Για να αποφύγουμε προβλήματα, η ΕΕ και η Νορβηγία αποφάσισαν να εναρμονίσουν τα τεχνικά μέτρα και την τρέχουσα νομοθεσία, τα νομοθετικά μέτρα στο μέγιστο βαθμό. Και σε μια ένα μέρος όπου η νέα νομοθεσία είναι διαφορετική από την νορβηγική νομοθεσία, ο τομέας αυτός αφορά τις απορρίψεις ηχθείων. Μέχρι σήμερα απαγορεύεται η απόρριψη πολλών ε, ειδών ε, από τέτοια αλλιεύματα και λέγεται ότι οποιοδήποτε αλλιέας, ε, οποιοδήποτε αλλιεύμα αλλιεύεται σε νορβηγικά χωρικά ύδατα πρέπει να εκφορτώνεται εκεί και αυτό από ό,τι γνωρίζετε είναι ασύμβατο με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί μικρότερου μεγέθους ηχθείες από αυτούς που επιτρέπεται να αλλιεύονται ή πέρα από τα επιτρεπόμενα αλλιεύματα πρέπει να εκφορτώνονται τα σκάφη μας θα έχουν προβλήματα λοιπόν όταν θα αλλιεύουν μέσα ε, στη, στα πλαίσια των χωρικών υδάτων της Νορβηγίας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο αποκτά κατεπήγοντα χαρακτήρα πλέον σήμερα η ΕΕ και η Νορβηγία συμφώνησαν να δημιουργηθεί μια τεχνική ομάδα για την προπαρασκευή και συζήτηση αυτών των ε, ε, προβλημάτων καθώς επίσης και των παράπλευρων αλλιευμάτων. Ε, σε σχέση με αυτή την ομάδα ε, τεχνικού χαρακτήρα που συμμετέχουν σε αυτήν ε, οι εκπρόσωποι των αλλιευτικών, των επιχειρηματιών, των αλλιέων και που παρουσίασε την έκθεσή της με βάση αυτά τα στοιχεία υπέβαλε την παρούσα της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πραγματικά δηλαδή μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, περιφερειοποιημένη προσέγγιση. η άμεσα εμπλεκόμενη του τομέα συνεργάστηκαν για να ταυτοποιήσουν και εντοπίσουν εκείνα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν η πρόταση που έχουμε παρουσιάσει έχει απαγόρευση απόρριψης αλλιευμάτων στο Σκάγκερακ. Μάλιστα και πριν από την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Το κάναμε αυτό ακριβώς επειδή ο στόχος και η πρόθεσή μας είναι να επιλύσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο απορρέει από την κατάργηση της Συμφωνίας Αλίας στο Σκάγκερακα. Χωρίς αυτή την συμφωνία για την απαγόρευση αυτών των απορριμμάτων, της απόρριψης αλλιευμάτων θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσουν να αλλιεύουν αλλιείς σε αυτή την περιοχή του Σκάγκερακ. Επαναλαμβάνω, αυτή η πρόταση δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο ως δεδομένο για την μεταρρύθμιση. Θα είναι απλά η κατάσταση ότι ένα πρόβλημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί και αυτή θα είναι η κατάσταση η οποία θα, όπως θα διαμορφωθεί θα μας δώσει μια ευκαιρία να αποκομίσουμε νέα νέα, μια νέα εμπειρία που θα είναι χρήσιμη στο πλαίσιο της αλληλευτικής μεταρρύθμισης. Επιτρέψτε μου να εισαγάγω τώρα σύντομα τα κυριότερα σημεία που εμπεριέχει αυτή η πρόταση. Πρώτον, στην πρόταση αυτή, στο άρθρο, το πρώτο, έχουμε την υποχρέωση να εκφορτώνονται όλα τα αλλιεύματα. Υποχρέωση να εκφορτώνονται όλα τα είδη τα οποία αναφέρονται στο παράτημα. Δεν είναι τα είδη. Για τα οποία προβλέπουμε απαγόρευση σε δύο κλίμακες. Προβλέπουμε απαγόρευση σε δύο κλίμακες. Προτείνουμε απαγόρευση των απορρίψεων μόλις τεθεί ε, σε ισχύ ο κανονισμός ε, για την πρώτη κατηγορία και μετά έχουμε μια δεύτερη φάση που θα τεθεί σε ισχύ δύο ε, χρόνια αργότερα η απαγόρευση. Τώρα θα πρέπει να εκφορτώνονται όλα τα αλλιεύματα τα οποία χρησιμοποιούν κάτω των 32 mm μάτι διχτυού. Και εξαίρεση θα υπάρξει μόνο για συγκεκριμένα είδη. Σε αυτή την πρόταση βασιζόμαστε στην κατάσταση λοιπόν των ειδών και στην προσέγγιση αλληλευτικής δραστηριότητας για το ΠΟΤ και το κρίλ. Δηλαδή να ε, εξαιρεθεί ο κιούρτος ουσιαστικά επειδή μπορεί το ψάρι να παραμείνει ζωντανό, πιάνεται ζωντανό. Στο άρθρο 4 έχουμε την υποχρέωση τα σκάφη να έχουν ε, επαρκείς ποσοστώσεις για όλα τα είδη. Όταν δεν υπάρχει πλέον ποσόσταση για κάποιο είδος, το οποίο υπόκειται στην απαγόρευση της απόρριψης, θα πρέπει να επανέρχεται στο λιμάνι το σκάφος. Άρα τα σκάφη θα πρέπει να οργανωθούν κατά τρόπον ώστε να έχουν τις ποσοστώσεις που θα τους δίνουν δυνατότητα να αλλιεύουν τα ίδια τα οποία βγαίνουν ε, στη θάλασσα. Το άρθρο 5 έχει να κάνει με τους γόνους. Ε, επομένως, δεν μπορούν γόνοι να πολλούνται προς ανθρώπινη κατανάλωση, εάν είναι κάτω δηλαδή από το επιτρεπόμενο μέγεθος. Ε, μόνο για φατρικούς σκοπούς θα μπορούσε να γίνεται κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει το ελάχιστο ε, μέγεθος της για το ψάρι που θα εκφορτώνεται, απλά επιτρέπεται η έγκαιρη, η γρήγορη προσαρμογή σε περίπτωση που χρειαστεί. Πάντα βέβαια αφού προηγηθεί επιστημονική εντολή. Το άρθρο 6 τώρα αφορά την εξειδίκευση των ελευτικών εργαλείων και εισάγει τεχνικά μέτρα τα οποία από κοινά έχουν συμφωνηθεί με την Νορβηγία για την μεγαλύτερη επιλεξιμότητα. Παράγραφος 3 του άρθρου αυτού έχει ως στόχο να επιτρέψει την γρήγορη εισαγωγή άλλων εργαλείων που έχουν είτε την ίδια είτε και καλύτερη ακόμη επιλεξιμότητα. Άρα έχουμε εισαγάγει την ευελιξία για να μπορούμε να καταλήξουμε σε πιο επιλέξιμα μέτρα. Μέτρα που θα, μάλλον σε εργαλεία τα οποία θα έχουν τη μεγαλύτερη επιλεξιμότητα. Στο άρθρο 7 λέμε ένα δίκτυ. Vessels can use just one gear. Ένα ε, σκάφος μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο μία κατηγορία δικτύου δηλαδή και όχι παραπάνω. Οι άλλε θα πρέπει να είναι αποθηκευμένε πάνω στο σκάφο. Το άρθρο 8 ξεκαθαρίζει ότι τα σκάφη που απορρίπτουν ε, ψάρια στη διάρκεια της παραμονής στο στη θάλασσα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες. Παραδείγματο χάρη, αν ένα σκάφος ξεκινήσει στο Σκάγκερακ και μετά περάσει στη Βόρεια Θάλασσα, ισχύουν γι' αυτό οι ίδιοι κανόνες και στη Βόρεια Θάλασσα. Εάν ξεκινάει το ταξίδι του στη Βόρεια Θάλασσα και δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό, τότε δεν επιτρέπεται να ψαρέψει ο Σκάγκερακ στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Κεφάλαιο 3 της πρότασης. Εισαγάγει τα μέτρα ελέγχου που έχουν συμφωνηθεί με την Ορβηγία. Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο σημείο που αναφέρεται στο άρθρο 11 και θα αποτελεί υποχρέωση για τα σκάφη κάτω των 50 μέτρων να είναι εξοπλισμένα με συγκεκριμένο εξοπλισμό μετά το 2014 θα ισχύει για όλα τα σκάφη μακρύτερα των 12 μέτρων από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Στο άρθρο 12 ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να καθιερώσουν ε, εθνικά μέτρα ελέγχου και επιθεωρήσεων που θα πρέπει να εισαχθούν στα εθνικά προγράμματα έλεγχου τους ώστε να επιτρέπει σε περίπτωση εξαιρέσεων ή νέων μέτρων να διασφαλίζεται ο έλεγχος των απορρίψεων και φυσικά αυτά τα νέα μέτρα θα πρέπει να ισχύουν. Η πρόταση περιλάμβανε κάποια τροποποίηση στην εξαίρεση. Θα αναφέρω δύο. Η πρώτη είναι ότι τα σκάφη που θα καλύπτονται από τον τρέχοντα κανονισμό εξαιρούνται από το καθεστώς προσπάθειας. Το δεύτερο, η δεύτερη, ε, ότι στην εξαίρεση θα αναγνωρίζεται ευελιξία 25% το πρώτο έτος και 15% το δεύτερο έτος και 10% στη συνέχεια για όλα τα είδη που καλύπτονται από την απαγόρευση απορρίψεων. Φυσικά μετά από αίτημα του τομέα προβλέπουμε μια ευελιξία ετήσιας ποσόστοση ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε από αυτή τη διαδικασία κάτι διότι θα είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζουμε κάποια τέτοια απαγόρευση απορρίψεων. Θα μάθουμε λοιπόν πολλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, τόσο εμεί όσο η διοίκηση και τα σκάφη. Σύμφωνα με την νομοθετική δομή, η δυναμή της συνθήκης της Έχουμε κάποια διάταξη για τις κατεξουσιοδότητες και τις εκτελεστικές πράξεις. Έτσι δίνεται εξουσία στην Κομισιόν να υιοθετεί κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις όπως αρμόζει. Για να προσαρμοζόμαστε στις τεχνικές και επιστημονικές προόδους χρονικά με αναλογικό τρόπο και για να εξασφαλίζουμε την απαραίτητη ευελιξία σε αυτές τις περιπτώσεις η Κομισιόν έχει προβλέψει ότι μπορεί να υιοθετήσει κατεξουδότηση πράξης για ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της πρότασης, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα τροποποίησης της διάταξης που σχετίζεται με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλλιευμάτων καθώς και τις διάταξεις που αφορά τις προδιαγραφές συγκεκριμένων εξοπλισμών και εργαλείων επιλεκτικότητας. Όπως ανέφερα, θα μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας Έχουμε προβλέψει λοιπόν κάποια μέτρα που θα μας επιτρέψουν σε όλους να καταγράψουμε και να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προσαρμόζουμε τους διάφορους κανόνες που προβλέπονται σε αυτή την πρόταση. Προς την ίδια κατεύθυνση έχουμε προτείνει την υιοθέτηση εκτελεστικών πράξεων για τον καθορισμό ε, επίπεδου εξοπλισμών, για παράδειγμα τις ελάχιστες απαιτήσει για ε, απομακρυσμένη παρακολούθηση των σκαφών. Τώρα, όπως εξήγησα στην αρχή, η οθέτηση αυτής της ε, πρότασης είναι επίγουσα. Ενθαρρύνουμε λοιπόν την Επιτροπή αυτή να συνεχίσει τις ε, συζητήσεις καθώς και το Συμβούλιο να επιταχύνουν τις συζητήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο Δεν έχουμε συμφωνία με την Νορβηγία Αυτό δεν είναι... που θα συνεχίσει να επιτρέπει. Έχουμε μόνο συμφωνία που θα επιτρέ... συνεχίσει να επιτρέπει τα δικά μα αλληλευτικά σκάφη να αλλιεύουν μέχρι την 1η Νοεμβρίου και πρέπει να δούμε τι θα γίνει αργότερα. Για τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αλλιεύουν σε νορβηγικά ύδατα. Αυτή η πρόταση λοιπόν θα μα επιτρέψει να καθιερώσουμε του κανόνε και έτσι τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να αλλιεύουν και να αποφύγουν τα προβλήματα ελέγχων και τήρηση των διαφορών κανόνων, των διαφορετικών κανόνων όταν αλλιεύουν σε νορβηγικά ύδατα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κούν, ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στο κέντρο μέσα σε αυτή τη συζήτηση εδώ και ένα εξάμεινο για την κοινή αλληλευτική πολιτική και βλέπουμε ότι η απόρριψη ηχθείων έχει κέρια σημασία ως πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Από το 2010 υπάρχει αυτή η ομάδα εργασίας ήδη για τον Σκάγκερακ μεταξύ της ΕΕ, δηλαδή Δανίας και Σουηδίας, από την Νορβηγία και δοκιμάζουν, ας το πω έτσι, τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης αλλιευμάτων. Πράγμα το οποίο είναι μια θετική διατύπωση κατεφημισμών της απαγόρευσης ε, εκφόρτωσης ε, παράπλευρων αλλιευμάτων ή σύλληψης παράπλευρων αλλιευμάτων. Και έχουμε εδώ τώρα τέτοια μέτρα που δεν υπάρχει καμιά ευκαιρία για το Ευρωκοινοβούλιο να εγκρίνει και πρέπει να εγκρίνει και το Συμβούλιο συνέχεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Είναι εις βάρος του Κοινοβουλίου. Προδικάζει αυτά που θα συμβούν στο μέλλον όσον αφορά την απαγόρευση για τέτοιου είδους παράπλευρα αλλιεύματα και τα, την εκφόρτωση αλλιευμάτων. Και όλα αυτά θα προδικάσουν το τι θα προταθεί στο μέλλον και τι θα ισχύει ως ρύθμιση. Γι' αυτό στο τέλος τέλος ε, υποχρεωνόμαστε να έχουμε επιτήρηση με βιντεοκυκλώματα, κυκλά, ε, κλειστά κυκλώματα των αλλιευτικών δραστηριοτήτων με τα 15, ε, για σκάφη 15 μέτρων και μεγαλύτερα και από το 2015 για σκάφη 12 μέτρων και μεγαλύτερα όταν δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιφέρεια. Και μετά όταν από, εξέρχονται από αυτή την περιφέρεια ε, αυτά τα μέτρα θα ισχύουν. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ προβληματικά όλα αυτά, διότι δεν έχουν αποσαφενιστεί πολλά πράγματα. Ποιος θα καθορίζει ποιες, ποια είδη έχουν μεγάλη πιθανότητα επιβίωσης. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την εποχή αλληλείας και τον εξοπλισμό αλληλείας. Όσον αφορά τώρα την επιλογή μεγέθους ηχθείων, ειδών ηχθείων, Όλα αυτά είναι επιβαρυντικά στοιχεία. Έχουμε ένα κατάλογο 30-40 ειδών ηχθείων στο παράτημα και αναφέρεται ότι από το 2013 απαγορεύεται η απόρριψη αυτών των αλλιευμάτων και το 2014 και εφ' απαγορεύεται η αλλίευση. Ποσοστώσεις λοιπόν, τι θα γίνει με, τη, ε, με τις ποσοστώσεις. Ελαστικότητα λέει 25% όσον αφορά αυτά τα αλλιεύματα για τα σκάφη το επόμενο έτος 15% μείωση, το επόμενο μεθεπόμενο έτος 10%. Αυτό είναι μια θετική προσέγγιση θα έλεγα. Πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε ότι είναι σωστό αυτό για τα ψάρια με τέτοιου είδους αλλιεύματα να μπορέσουν να είναι βιώσιμα ώστε με την ε, ε, αλλίευσή τους να μπορούμε να έχουμε ας το πω έτσι ε, μια θετική κατάσταση. Αυτά είναι πολλά πράγματα τα οποία από κοινού πρέπει να συζητηθούν μικρότερα σκάφη έχουν δυσανάλογες δαπάνες. Οι τα μεγάλα σκάφη μπορεί πιο εύκολα να λειτουργούν εκεί τα πράγματα. Οι μηχανισμοί ελέγχων όμως που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηλεκτρονικού χαρακτήρα και έχουν διευρυνθεί στην ηλεκτρονική συνιστόσα. Κάθε σκάφος όταν φεύγει από το λιμάνι και πάει να αλλιεύσει πρέπει να, να το αναφέρει αυτό στην αρμόδια αρχή Μέσω του IES υπάρχει αυτόματα το σύστημα εντοπισμού, αυτόματο εντοπισμού του σκάφους. Η ηλεκτρονική επαγρύπνηση, με ποια ταχύτητα ε, κινείται αυτό ε, το σκάφος, πότε φτάνει στο χώρο αλίευσης, ε, τι κάνει με τη... Οι χώροι αλίευσης είναι γνωστοί, δύο ώρες πιο πριν πρέπει να γνωστοποιεί στην αρχή στον ελεγκτικό οργανισμό αυτής αρμόδια χώρα ότι πάει να λιεύσει εκεί τα λοιπά Μία, ας το πω έτσι, βίντεο επιτήρηση είναι ο μεγάλος αδερφός πλέον, το καθεστώς του μεγάλου αδερφού και αυτό είναι απόλυτα πραγματικά καταχρηστικό και υπερβολικό. Πρέπει να έχουμε χρόνο και όλα αυτά να τα συζητήσουμε επαρκώς, διότι όταν έχουμε ένα τέτοιο κανονισμό, ε, αυτά θα ισχύουν ε, σε σχέση με την κοινή αλλιευτική πολιτική και θα τα έχουμε όλα αυτά μπροστά μας Δηλαδή αν όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν έτσι, γιατί να μην λειτουργούν ε, παντού με τον ίδιο τρόπο. Πολύ βιαστικά κινούμαστε νομίζω. Οι σκιώδεις εισηγητές πρέπει και αυτοί να δραστηριοποιηθούν. Πρέπει να έχουμε χρόνο και με τους εκπροσώπους των ε, ψαράδων των αλλιέων στα κράτη μας να συζητήσουμε πόσο αυτά επηρεάζουν, οι απόψεις τους μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα. Με πολύ κριτικό και επικριτικό πνεύμα αντιμετωπίζω αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Øh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα πώς είπα μόλις πριν ο κύριος Κούν. Φυσικά και εγώ στηρίζω την ιδέα αυτού του πιλωτικού σχεδίου για την απαγόρευση των απορρίψεων. Είναι μια καλοδεχούμενη πρόταση, αλλά είναι και μια πρόκληση να είναι έτοιμα όλα μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Περί αυτού ε, πρόκειται, αφού τότε λύγει η τρέφουσα συμφωνία. Και για την 1η Ιανουαρίου πάλι θα ήταν δύσκολο βέβαια. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πιστεύω ότι απαιτούν περαιτέρω διευκρίνηση και δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνος στη διάθεσή μας. Θα εστιάσω τώρα λοιπόν ε, στα ερωτήματά μου. Και όταν η Επιτροπή τονίζει ότι δεν πρόκειται αυτό να αποτελέσει προηγούμενο για άλλους τομείς, αλλά ότι θα εφαρμόζεται μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εγώ αγχώνομαι και ξέρω ότι αγχώνεται και η βιομηχανία για το κατά πόσον αυτό αληθεύει. Γιατί είναι δύσκολο μεν να υιοθετήσει μια τέτοια ε, διάταξη, αλλά μετά εύκολο να την μεταφέρει και σε άλλου τομεί. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υποτιμήσουμε το ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία η αλής, η βιομηχανία. Και κάποια πράγματα στην αλληλευτική μας πολιτική εν γέννη δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε. Μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Μην αφήσουμε εκτός τους κατεξοχήν ενδιαφερόμενους και γνώστες. Είπατε ότι έχει συγκροτηθεί μια ομάδα εργασία για αυτά τα ζητήματα και είναι πολύ επικοδομητικό και έχει συγκροτηθεί από κάτω προς τα πάνω. Το ερώτημά μου είναι όμως μέχρι στιγμής σε αυτήν την ομάδα εργασίας ποιος συμμετείχε και γιατί εμείς δεν είδαμε μια ανάλυση, ε, μια μελέτη του αντικτύπου μετά από την υιοθέτηση αυτής της απαγόρευσης απορρίψεων για το Σκάγκερακ, εφόσον αυτό ισχύσει, γιατί αυτό θα επηρεάσει πολλά κράτη-μέλη και όχι μόνο αυτά στα οποία αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Βρετανία και αυτά τα κράτη εμπλέκονται. Έχετε έρθει σε επαφή με αυτά τα κράτη και τι έχουν να πούν για αυτή την απαγόρευση. Τώρα, όπως έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να είμαστε πλήρως, ε, πρέπει να έχουμε την πλήρη ε, ενημέρωση και αυτό πρέπει να γίνεται με επιτήρηση μέσω κάμερας. Λέτε ότι πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση, αλλά αν τα νορβηγικά σκάφη δεν έχουν αυτά τα συστήματα, εντάξει δεν είναι μέλος της Ένωσης, αλλά δεν θα έπρεπε και αυτά να τηρούν αυτές τις ε, υποχρεώσεις. Και τι επιπτώσεις θα υπήρχαν εάν ενεκρίνονται ο προτάσεις αυτές. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει απαγόρευση της αλίας ως κάγκερακ. Πάντως θα συνεργαστώ με τα χαράς και με τον εισηγητή και με τους κοιόδες γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση και θέλω να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι δεν είναι ένας τομέας που εγώ θέλω να ε, υποστηρίξω του αλείς απλά και μόνο είναι ένας ε, τομέας που εντάσσεται στην κοινή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριε, κύριε είναι η κυρία Λόβιν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με την απαγόρευση εδώ και 30 χρόνια από το 1980 στην Νορβηγία της απόρριψης παράπλευρων αλλιευμάτων είναι σαφές εδώ ότι έχουμε ένα πρόβλημα εφαρμογής. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων με την Νορβηγία όταν δραστηριοποιούνται σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χωρικά ύδατα της Νορβηγίας. Το βρίσκω εξαιρετικό για το ότι η Νορβηγία, η Σουηδία και η Δανία ως καλοί γείτονες κατάφεραν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και κατάφεραν από πλευρά κυβερνήσεών του να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση. Θέλουμε εδώ να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απαγόρευση ε, απόρριψη αλλιευμάτων για τον κύριο Κούν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέπεται κανείς να είναι προπομπό ή πρωτοπόρο ως χώρα στην παγκόσμια νομοθεσία με την λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Όταν κάποιο προσπαθεί να αλλιεύσει θα μπορεί να είναι καλύτερος μέσα σε ένα αυστηρότερο, αυστηροποιημένο ε, πλαίσιο. Και θα ήθελα σε σχέση με ε, την συνάδελφο να πω ότι για αυτές τις τρεις όμορες χώρες μπορούν να δείξουν ότι είναι πρωτοπόρες και για την εισαγωγή της απαγόρευσης ε, ε, απόρριψης ε, παράπλευρων αλλιευμάτων λέγεται ότι είναι δύσκολο λέει να επαληθεύεται αυτό η Νορβηγία κατέδειξε ότι είναι βιώσιμο και μπορεί να, να αναφερθεί ότι είναι μια βιώσιμη πορεία μια θετική οδός αυτή. Έχω κάποια σημεία στα οποία με επικριτικό πνεύμα αντιμετωπίζω τα, κάποια στοιχεία της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόρριψη, ε, για παράδειγμα, τα απορριπτόμενα αλλιεύματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς και ε, για τέτοια χρήση. Θα ήθελα να πω ότι το θεωρώ λανθασμένο να δημιουργηθεί μια αγορά στην οποία θα διοχετεύονται αυτά τα προϊόντα των παράπλευρων αλλιευμάτων σε σχέση με τη Δανία, την ε, Σουηδία, Νορβηγία μπορεί ίσως αυτό να θεωρείται δεδομένο υπό αυτό το πλαίσιο. Σε άλλες χώρες όμως θα ήταν ε, αναγκαίο για συσίτια να δούμε την ανάγκη διάθεσης τέτοιων ε, αλλιευμάτων που δεν μπορούν να διατεθούν αλλού, αλλά είναι μια ολιστηρή πορεία αυτή. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι για το τι μπορεί να αλλάξει με βάση επιστημονικά τεκμήρια και στοιχεία πρέπει να δρούμε και πάντα με βάση την, ε, τα επιστημονικά αυτά, ε, τις επιστημονικές συστάσεις έχουμε τα μάτια των δικτυών που είναι πλέον ε, μικρά για να μην μπορούν να συλληφθούν γόνοι και προτού έχουν οριμάσει τα ε, ψάρια, προτού έχουν ενηλικιωθεί τα ψάρια. Θα ήθελα να ακούσω ποιε είναι οι απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτέ τι ε, ε, συνιστώσει. Υπάρχουν είδη τα οποία μπορούν να αλλιεύονται από την άλλη πλευρά. Έχουμε τον μπακαλιάρο για παράδειγμα. Έχουμε και τα καβούρια που πολλές φορές στο ίδιο δίχτυ ως αλλιεύματα συλλαμβάνονται και ε, φτάνουν στο κατάστρωμα ενός ε, ψαράδικου. Ε, υπάρχουν και άλλα ψάρια τα οποία ως ε, παράπλευρα σύνθετα σε ένα μεικτό αλίευμα μπορούν να εντοπίζονται. Δύο ίσως ειδών ψάρια, τρία είδη ψάρια, ψαριών στο ίδιο δίχτυ. Το θέμα των ελέγχων λοιπόν. Εδώ αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε κάποια σημεία αναφοράς για το στόλο μας Λοιπόν, έχουμε αποτελέσματα θετικά και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παράπλευρων αλλιευμάτων. Όταν λειτουργεί, ε, έχουμε ένα κανονικό ε, εξοπλισμό, μπορούμε να δούμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα καλά και μπορούμε αμέσως να ε, διαπιστώσουμε αν κάτι δεν πάει καλά και αν υπάρχουν προβλήματα με παράπλευρα αλλιεύματα. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όπως πιστεύει κάποιος καμιά φορά. Ευχαριστώ. Κυρία Φράγα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς την ε, Επιτροπή στον κύριο ε, Κούν. Αν μπορεί να απαντήσει. Αυτά τα τεχνικά μέτρα θα ενταχθούν στο πλαίσιο μιας διεθνής αλληλευτικής συμφωνίας. Τι εννοώ. Πιο πολύ το λέω για την νομική βάση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια διεθνής αλληλευτική συμφωνία για αυτά. Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε εσείς εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, συμφωνώ μάλλον με τον εισηγητή. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο προβληματισμού και προετοιμασίας. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι ήταν πολύ δύσκολη δουλειά και για την Κομισιόν, για όσους ενεπλάκησαν σε βάθος σε αυτή την άσκηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πρέπει να πω ότι η Νορβηγία μας κατάπληξε όλους ε, ανακαλώντας τη συμφωνία της και πράγματι οι τρεις χώρες η Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία, και, καθώς και η Γερμανία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, αμέσως ε, χρησιμοποίησαν πολιτικές διατάξεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και ήδη τον περασμένο Ιανουάριο προέβησαν σε δήλωση όπου δεσμεύτηκαν πολιτικά για να προτείνουν απαγόρευση απορρίψεων για το Σκάγκερακ. Ήταν λοιπόν πολύ εντατικέ οι εργασίε από τεχνική άποψη για να μπορέσουν να προσδιοριστούν όλα τα μέτρα που αρμόζουν και που περιλαμβάνονται πλέον σε αυτόν τον κανονισμό. Ήθελα να υπογραμμίσω όπως ε, αναφέρθηκε θελήσαμε να κάνουμε αυτή την εργασία σε τεχνικό επίπεδο το οποίο σημαίνει ότι υπήρξε μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν όχι μόνο διοικητικοί υπάλληλοι αλλά και εκπρόσωποι της βιομηχανίας, δηλαδή αυτοί που θα υλοποιήσουν τα εν λόγω μέτρα. Συμμετείχαν επίσης ε, και ΜΚΟ που συνεργάστηκαν όλοι αυτοί μαζί σε τεχνικό επίπεδο για να προσδιορίσουν τόσο τα είδη όσο και τα τεχνικά μέτρα όσο και τα μέτρα ελέγχου. Ήταν λοιπόν πολύ εντατικέ, ε, δύσκολε εργασίε σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για να φτάσουμε στην ε, διαμόρφωση αυτή τη πρόταση. Τώρα λοιπόν ήθελα να υπογραμμίσω ότι πράγματι δεν προκαταβάλει τις συζητήσεις των μεταρρυθμίσεων αυτή η πρόταση. Τις προβλέπει, όπως προβλέπει και την περιφερειοποίηση, δηλαδή παρέχει τη δυνατότητα σε διοικήσεις, κράτη, σε τομείς που πρώτοι θα επηρεαστούν από ορισμένα νούμερα να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να μπορέσουν να υιοθετήσουν τα μέτρα εκείνα που είναι σημαντικά για αυτούς. Αυτή η πρόταση λοιπόν προβλέπει κατά κάποιο τρόπο την περιφερειοποίηση. Προβλέπει κατά κάποιο τρόπο τη νέα πολιτική για την απαγόρευση απορρίψεων, αλλά δεν προκαταβάλει τις μελλοντικέ συζητήσεις, διότι είναι κάτι που θα εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τομέα μόνο. Αντιθέτως, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μάθουμε τι σημαίνει πραγματικά η υλοποίηση συγκεκριμένα αυτών των νέων κανόνων. Θα είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε εμπειρικά πλέον ε, πάνω στην υλοποίηση πρόκειται για ένα είδος πιλωτικό έργο. Θα μας επιτρέψει να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι πραγματικές δυσκολίες όταν λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά τα πράγματα και ποιες δυσκολίες πρέπει να λάβουμε υπόψη για τις ε, συζητήσεις μας στο μέλλον. Έτσι λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι να μελετήσουμε τις διάφορες προτάσεις και συστάσεις ε, που θα μας γίνουν για συγκεκριμένες πτυχές της μεταρρύθμισης. Ποια θα είναι η αντίδραση της Νορβηγίας εάν πράγματι τα μέτρα δεν υιοθετηθούν τάχιστα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Φυσικά έχουμε επισημάνει στην Νορβηγία σε όλα τα πολιτικά επίπεδα ότι η διαδικασία εγκρισής μας, υιοθέτησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο. Προς το παρόν το μόνο που έχουμε πετύχει είναι να έχουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κύριων ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα από τώρα μέχρι την 1η Ανδρίου και στο μεταξύ προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τους συνομιλητές μας για να αναγνωρίσουμε τα μέτρα που θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εν αναμονή της ε, υιοθέτησης αυτής της πρότασης. Ε, παρ' όλα αυτά, φυσικά, τα λιευτικά σκάφη που αλλιεύουν στην περιοχή θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, πραγματικά, συγκεκριμένα ή θα συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με την Νορβηγική νομοθεσία. Δεν μπορούν να συμμορφώνονται και με τις δύο νομοθεσίες. Έτσι λοιπόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ήθελα να υπογραμμίσω τα στοιχεία προβληματισμού που σχετιζόνται με το πώς θα πρέπει να πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα αλλιεύματα που θα εκφορτωθούν. Τώρα εφαρμοστέ στο η δυνατότητα χρήση των αλλιευμάτων που κανονικά θα απορρίπτονταν να χρησιμοποιηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο τρόπος, αυτή η πρόταση αποφυγής οποιοδήποτε κέρδους που θα μπορούσε να αλλοιώσει, να διαστρεβλώσει τη λειτουργία της αγοράς, που θα μπορούσε να ε, δώσει κίνητρα για μη απορρίψεις με σκοπό οποιοδήποτε, οποιασδήποτε μορφής κέρδος. Η συζήτηση λοιπόν για το τι θα γίνεται με τις απορρίψεις των αλλιευμάτων που εκφορτώνονται μπορεί να αποτελέσει ένα ζήτημα. Όσον αφορά το σχόλιο για τα τεχνικά μέτρα που και τη σκέψη αυτή μιας διεθνούς συμφωνίας, αυτά είναι τα τεχνικά μέτρα που είναι απαραίτητα για τα ευρωπαϊκά σκάφη. Σκόπος λοιπόν του κανονισμού είναι να προβλέψει όλες τις προσαρμογές, όλες τις εξαιρέσεις στον κανονισμό στα τεχνικά μέτρα που είναι απαραίτητες ώστε να επιτρεπεί νομιμότατα στα σκάφη να αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή. Όσον αφορά το αντίκτυπο αυτών των προτάσεων. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι πράγματι δεν έχει γίνει εκτίμηση δικτύπου διότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου μεταφέραμε στην ευρωπαϊκή μας νομοθεσία τις συνέπειες διεθνών συμφωνιών ή ανάκλησης διεθνών συμφωνιών εκ μέρους μιας τρίτης χώρας. δηλαδή δεν προλάβαμε ούτε υπήρχαν οι συνθήκες οι κατάλληλε ώστε να μπορέσουμε να προβούμε σε εκτίμηση αντικτύπου των προτινόμενων μέτρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και το σημείο αυτό. Σημείο 14 της διάταξη, διάταξης, επόμενη συνεδρίαση. Α, όχι, στα διάφορα δεν υπάρχει τίποτα. Και 16 ανακοινώσει του Πρόεδρου σχετικά με τι αποφάσει που έλαβαν οι συντονιστέ. Τι είπαμε το πρωί, ποιε είναι οι συστάσει τι γνωρίζετε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνονται. Επόμενη συνεδρίαση λοιπόν 8 Οκτωβρίου το απόγευμα και 9 Οκτωβρίου πρωί και απόγευμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σα ευχαριστώ όλου για την παρουσία σα, την εργασία σα και τι ερμηνεί. Ε,